Okay. Can I have your attention, please? Παρακαλώ. We are starting... Αρχίζουμε τη δεύτερη, το δεύτερο τμήμα του σεμιναρίου για τους δημοσιογράφους. Σήμερα θα αρχίσουμε με την παρουσιάσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του επόπτη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα μιλήσει ο κύριος Ριχάρδος Σόστακ που είναι μέλος του γραφείου της κυρίας Ρέντινγκ, της Επιτρόπου Ρέντινγκ και που χειρίζεται ένα από αυτά τα βασικά θέματα με τα οποία ασχολείται η κυρία Ρέντινγκ. Επίσης έχουμε από την Υπηρεσία Επιτήρησης των Προσωπικών Δεδομένων, τον κύριο Χάιμερς, που είναι υπεύθυνο για τις νομοθετικές γνωμοδοτήσεις που είναι και αυτό από τα κυριότερα θέματα που αφορούν την νομοθεσία και την προσεχή οδηγία. Πρώτα λοιπόν θα μιλήσει ο κύριος Ρίτσαρτ Σόστακ. Καλημέρα. Good morning to everybody. So I've been invited to speak a little bit about the... Θέλω να σας μιλήσω λίγο για την προοπτική που έχει η Κομισιόν για το μεταρρυθμιστικό πακέτο ή δέσμη για την προστασία των δεδομένων. Όπως ξέρετε προτείνουμε και κανονισμό και οδηγία και θα ξέρετε κι εσείς από τις συζητήσεις σας τα βασικά. Οι κύριες ιδέες της Κομισιόν είναι το θέμα μου για να καταλάβετε γιατί υποβάλλονται οι προτάσεις αυτές και ποιοι είναι οι στόχοι τους. Αρχίζω λοιπόν με την ισχύουσα κατάσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη και μερικά από τα προβλήματα που θέλουμε να λύσουμε. Ισχύει μια οδηγία από το 1995, δηλαδή έχουν ήδη υπάρξει κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από το 1995 στην Ευρώπη. Εδώ και 18 χρόνια δηλαδή. Αυτό είναι η αφετηρία. Μπορεί να έχετε ακούσει ότι η Κομισιόν ε, δεν προτείνει τίποτα το επαναστατικό, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα σημαντικό εδώ και 18 χρόνια. Αυτά όλα είναι λάθος. Το θέμα είναι ότι το 1995 Ε, είναι πολύ, κάτι που απέχει πολύ χρονικά. Τότε ήταν 11 τα μέρη, δεν υπήρχε το Google, δεν υπήρχαν τόσο κινητά, οι κεραίες ήταν ύψους 15 μέτρων και τέτοια πράγματα. Αυτά έχουν όλα αλλάξει και επομένως το θέμα δεν είναι αν είναι σημαντικός ή όχι ο ιδιωτικός χαρακτήρας ή αν χρειάζεται προστασία δεδομένων, αλλά απλώς εάν οι κανόνες που ισχύουν από το 1995 αρκούν και για σήμερα, αν έχουν νόημα ή αν χρειάζονται εξυγχρονισμό, ενημέρωση. Αυτό είναι η αφετηρία λοιπόν. Υπάρχουν κανόνες εδώ και το 1995 που λειτουργήσαν καλά μέχρι τώρα και που δημιούργησαν υψηλό επίπεδο προστασίας. Αυτό θέλουμε να εξετάσουμε. Δεύτερον, από το 1995 οδηγία ισχύει και το χαρακτηριστικό της μιας οδηγίας είναι ότι πρέπει να μεταφερθεί υποχρεωτικά στην εθνική νομοθεσία του κάθε κράτους. <clears throat> Υπάρχει δηλαδή ένα ενωσιακό νομοθέτημα που σε ακολουθείται από 25 και σε λίγο 28 ε, εθνικούς νόμους. Στη Γερμανία ας πούμε υπάρχουν 31 σημεία της οδηγίας αυτής που μεταφέρθηκαν σε 66 νομοθετικά σημεία στην εθνική νομοθεσία συν πρόσθετους νόμους για τα κάθε κρατήδιο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη δεν βασίζεται μόνο σε μία οδηγία του 95, αλλά και στα 66 γερμανικά νομοθετήματα πολλαπλασιασμένα επί τα υπόλοιπα κράτη. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται πολύπλοκα, γιατί καμιά φορά υπάρχει έλλειψη συνέπειας. Αυτή λοιπόν είναι η βάση. Από τη μία υπάρχει ήδη μια οδηγία που θεσπίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και από την άλλη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο, πολύπλοκο, πάρα πολύ πολύπλοκο σύστημα για τη μεταφορά στα κράτη-μέλη. Τι προσπαθούμε λοιπόν να πετύχουμε εμείς τώρα. Πρώτον, θέλουμε να δούμε τις περιπτώσεις όπου θέλουμε από την Κομισιόν να υπάρξει μεγάλη αλλαγή και μετά περιπτώσεις όπου δεν ζητούμε αλλαγή για να καταλάβετε λίγο τη δυναμική των πραγμάτων. Ποια είναι η κυριότερη αλλαγή λοιπόν που προσπαθούμε να πετύχουμε. Προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε μια οδηγία του 95 κείμενο δηλαδή που εφαρμόζεται διαφορετικά από το κάθε κράτος μέλος, σε έναν ενιαίο κανονισμό που να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλες τις χώρες μέλη. Όπως μία είναι η Ένωση, ένας θα είναι και ο σχετικός νόμος. Αντί για γερμανικό ομοσπονδιακό νόμο με 66 ρήτρε επί 27 χώρες μέλη, θέλουμε ένα νομοθέτημα. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτή είναι η κυριότερη και σημαντικότερη αλλαγή που προτείνουμε και προσπαθούμε να πετύχουμε. Γι' αυτό μπορεί να ακούτε καμιά φορά ότι ορισμένοι λένε ότι οι επιχειρηματίες δεν είναι ικανοποιημένοι κλπ. Αλλά αυτό το ότι δηλαδή θέλουμε να περάσουμε από 27 εθνικά νομοθετήματα σε ένα είναι κάτι το οποίο υποστηρίζεται πάρα πολύ και από τους επιχειρηματίες και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η δεύτερη αλλαγή που θέλουμε είναι η εξής. Αφού θα υπάρχει ένα ενιαίο νομοθέτημα, τότε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την Ένωση. Μια εταιρεία που δράσει και στις 27 χώρες μέλη, αυτή τη στιγμή πρέπει να εφαρμόζει 27 νομοθετήματα, τώρα θα χρειάζεται να αντιμετωπίσει και να εφαρμόσει μόνο ένα. Η εταιρεία λοιπόν θα γνωρίζει ποιος είναι ο ρυθμιστής και δεν θα χρειάζεται να αντιμετωπίσει 27 διαφορετικούς. Πρόκειται λοιπόν και για απλοποίηση και αυτό ικανοποιεί πολύ τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι λοιπόν η μεγαλύτερη και κυριότερη αλλαγή. Δεύτερη αλλαγή που προτείνουμε αφορά το θέμα της εφαρμογής. Θα έχετε ακούσει ότι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες έχουν πάρει συμβουλές για την καλύτερη προστασία αλλά δεν τις εφαρμόζουν. Άρα χρειάζεται καλύτερο συντονισμό των συντονιστικών αρχών ή εποπτικών αρχών. Ορισμένοι επόπτες έχουν πολύ περιορισμένες δικαιοδοσίες, άλλοι περισσότερες. Πολλοί δεν μπορούν καν να εφαρμόσουν ένα πρόστιμο στις εταιρείες που αραβιάζουν την νομοθεσία. Θέλουμε λοιπόν οι κανόνες που θα ισχύουν στην Ευρώπη να εφαρμόζονται κιόλα. Και αυτό θέλουμε να το πετύχουμε μέσω περισσότερων δικαιοδοσιών στους επόπτες ή στους υπεύθυνους για την προστασία των δεδομένων. Αυτές είναι οι δύο κύριες αλλαγές. Ένας ενιαίος νόμος για ολόκληρη την Ευρώπη και διασφάλιση της σωστής του εφαρμογής. Τώρα, πού δεν ζητούμε αλλαγές. Στην ουσία της νομοθεσίας. Στην ουσία στα δικαιώματα των ατόμων δηλαδή. Γιατί σας ξαναείπα, υπάρχει οδηγία από το 1995 που προβλέπει υψηλό επίπεδο προστασίας που έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Το θέμα όμως είναι αν είναι ενημερωμένοι οι κανόνες αυτοί, εξυγχρονισμένοι. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε επανάσταση, απλώς μια, έναν εξυγχρονισμό, μια προσαρμογή στα τωρινά δεδομένα. Δεν προτείνουμε λοιπόν μεγάλες αλλαγές στην ουσία, στο περιεχόμενο της νομοθεσίας. Τα δικαιώματα των ατόμων παραμένουν τα ίδια με μια απλή ενημέρωση. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Μπορεί να, ξέρετε, να έχετε ακούσει ότι για τη συγκατάθεση λέγονται πολλά. Πολλοί θεωρούν ότι η συγκατάθεση σημαίνει ότι κάθε φορά που ανοίγει τον υπολογιστή σας θα βγαίνει ένα παράθυρο που θα ζητάει η συγκατάθεση όποτε ζητάτε οτιδήποτε στο φιλομετρητή σας και ότι αυτό θα καταστήσει τα πράγματα πολύ δύσκολα και αδύνατα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν θα γίνεται έτσι η συγκατάθεση. Δεν θα ζητιέται έτσι η συγκατάθεση. Η συγκατάθεση είναι ένα από τα έξι κριτήρια που καθιστούν θεμητή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτείται συγκατάθεση, σε άλλες όχι. Παραδείγματος χάρη, αν υπογράψετε ένα συμβόλαιο όπου δίνεται συγκατάθεση, δεν ζητιέται και δεύτερη. Αν μια εταιρεία προβάλλει μια διαφήμιση στην οθόνη σας που βασίζεται σε προηγούμενες πληροφορίες από προηγούμενη σας φιλομέτρηση, χρειάζεται απαραίτητο συγκατάθεση και όχι, διότι Υπάρχουν άλλοι λόγοι όπως το θεμητό συμφέρον που επιτρέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση των ενδιαφερομένων. Είναι λίγο όπως τα αυτοκίνητα. Βάζετε τη δεύτερη ταχύτητα και αν θέλετε να πάτε πιο γρήγορα περνάτε στην τρίτη. Γιατί αλλιώς θα ζεσταθεί η μηχανή. Κάτι τέτοιο ισχύει και εδώ. Αν δεν είναι πολύ ενοχλητική η συγκατάθεση αν είναι πιο σημαντική χρειάζεται, παραδείγματος χάρη. Μία περίπτωση όπου δεν χρειάζεται συγκατάθεση. Η άμεση εμπορία. Θεωρούμε ότι απλώς είναι θεμητό για μια εταιρεία να σας στείλει μια διαφήμιση, καταρχήν γιατί την ωφελεί και από την άλλη γιατί δεν παραβιάζει τον ιδιωτικό χαρακτήρα των δικαιωμάτων Αν όμω είναι πιο σημαντική αυτή η παρεμβολή, τότε χρειάζεται συγκατάθεση. Δεν προτείνουμε καμιά αλλαγή εδώ. Το μόνο που κάνουμε είναι σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται, απαιτείται συγκατάθεση, που είναι οι ίδιες με αυτές που προέλεπε η οδηγία, τότε η, συγκατά... αίτηση συγκατάθεση να είναι ρητή και ασαφής γιατί αν θέλουμε να υπάρχει εμπιστοσύνη στον τρόπο λειτουργίας του ίντερνετ και θέλουμε να συνεχίσει ο κόσμος να αγοράζει από το ίντερνετ και άρα να χορηγεί προσωπικά δεδομένα, τότε η συγκατάθεση πρέπει να γίνεται με σαφή τρόπο και να είναι πραγματική και ρητή Δεν θα χρειάζεται συγκατάθεση σε όλες τις περιπτώσεις. Όποτε όμως χρειάζεται τότε πρέπει να είναι σαφής και ρητή η συγκατάθεση. Γιατί τα λέω λοιπόν αυτά, γιατί η πρόταση ότι με, την, με τον κανονισμό θα χρειάζονται σε περισσότερες περιπτώσεις συγκατάθεση δεν ισχύει. Εμείς λέμε απλώς ότι όπου χρειάζεται, όποτε χρειάζεται συγκατάθεση τότε να είναι πιο πραγματική η σιωπή δεν είναι το ίδιο πράγμα με την ρητή συγκατάθεση. Τώρα, το δικαίωμα στη λύθη. Και αυτό ακούγεται ότι θα αλλάξει τα πάντα. Όχι, όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ήδη υπάρχει στην ισχύουσα νομοθεσία που λέει ότι υπάρχει το δικαίωμα να σβηστεί κανείς από τον κατάλογο μιας εταιρείας. Όποτε δεν χρειάζονται τα δεδομένα σας πρέπει να σβήνονται. Το μόνο που αλλάζουμε ως προς αυτό είναι ότι λέμε ότι όταν κάποιος ζητάει από μια εταιρεία να σβήσει τα στοιχεία του, γιατί δεν χρειάζονται, τότε πρέπει να σβήνονται τα στοιχεία. Δηλαδή ο πολίτης έχει το δικαίωμα να πει θέλω να σβηστούν τα στοιχεία μου, τότε πρέπει να σβήνονται υποχρεωτικά, εκτός αν είναι απαραίτητο να κρατηθούν. Δεν αλλάζουμε λοιπόν την ισχύουσα νομοθεσία. Ούτε πρόκειται για τίποτα επαναστατικό ή καινούριο καινοτόμο. Είναι κάτι που ήδη προβλέπεται από την οδηγία του 95. Εμείς απλώς το ενδυναμώνουμε λιγάκι, το προσαρμόζουμε στην νέα ψηφιακή οικονομία, τίποτε παραπάνω. Το άλλο επιχείρημα που ακούγεται, και αν κάποιο στοιχείο κυκλοφορεί γενικά στο ίντερνετ και γίνεται δημόσιο, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση με τη λογική θα αντιδράσετε. Γνωρίζουμε ότι αν τα δεδομένα περάσουν στο ανοιχτό ίντερνετ δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα εκτός αν υπάρξουν νέες τεχνολογικές λύσεις. Το θέμα όμως είναι ότι αν μια εταιρεία μεταφέρει, πουλάει προσωπικά δεδομένα σε μια άλλη εταιρεία τότε υπάρχει χνηλασιμότητα και μπορεί να απαγορευτούν και να σβηστούν. Δεν ζητούμε τίποτα το αδύνατο δηλαδή. Απλώς ενδυναμώνουμε το δικαίωμα της διαγραφής. Εφόσον είναι γνωστή βέβαια η αλυσίδα της μεταφοράς. Ξέρω ότι εδώ υπάρχουν δημοσιογράφοι και το δικαίωμα αυτό στη διαγραφή δεν σημαίνει ότι μπορούμε να σβήσουμε οτιδήποτε γράφει μια εφημερίδα διαβάστε την οδηγία θα δείτε λέει ότι δεν αφορά θέματα προστασίας της ελευθερίας του λόγου. Δεν ζητάμε λοιπόν αλλαγή των κανόνων, τους προσαρμόζουμε απλώς στη σύγχρονη εποχή. Και τα επιχειρησιακά πρότυπα όπως λειτουργούν σήμερα δεν πρόκειται να αλλάξουν ούτε να υπονομευθούν. Κάτι άλλο που δεν αλλάζουμε είναι το πεδίο εφαρμογής. Η οδηγία του 1995 δεν αφορούσε την εφαρμογή του νόμου, αλλά μιλούσε για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Και αυτό είναι λογικό, γιατί ο δημόσιος τομέας μπορεί και αυτός να γνωρίσει περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και του απόρριτου. Ιδίως στον τομέα της υγείας, στα υγειονομικά στοιχεία. Και ο δεύτερος πιο ευαίσθητος τομέας είναι ο δημόσιος τομέας. Ίσως και γιατί εκεί τα υγειονομικά είναι κυρίως δημόσια. Έπειτα, οι γενικές αρχές της προστασίας των δεδομένων, δηλαδή να παραμένουν στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο κλπ. Ισχύουν και για τον ιδιωτικό και για το δημόσιο τομέα. Και τρίτον, δεν μπορεί να γίνει μια απόλυ... ένας απόλυτος διαχωρισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αν μια δημόσια αρχή θέλει για να μειώσει το κόστος της να, να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο του cloud, τι θα θεωρείται αυτό, δημόσιο ή ιδιωτικό. Ήδη και από την οδηγία του 95 αναφερόταν αυτά τα προβλήματα και ισχύουν και για σήμερα. Σε μερικές περιπτώσεις βέβαια οι δημόσιες αρχές μπορεί να χειριστούν ή να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα με δημόσιο τρόπο, αλλά Βασικά δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε. Αυτά είχα να σας πω. Και αν ήθελα να τα συνοψίσω θα έλεγα απλώς τα εξής τρία πράγματα. Ένα. Ήδη υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1995. Όταν λοιπόν σας πει, αν σας πει κάποιος ότι είναι οι κανόνες της Κομισιόν θα αλλάξουν άρδιν τα πράγματα, να μην το πιστέψετε. Να ρωτήσετε Είστε σίγουρος ότι είναι κάτι διαφορετικό από τα ισχύοντα. Δεύτερον, οι κύριες αλλαγές προβλέπουμε αφορούν τη δομή της προστασίας των δεδομένων, δηλαδή ένα ενιαίο νομοθέτημα και επιβάλλεται μεγαλύτερη επιβολή του νόμου. Και τρίτον, η ουσία των κανόνων είναι εξέλιξη και όχι επανάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Χίλκε Χάιμαντς. Ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω μερικά στοιχεία σε αυτά που μόλις σας είπε ο Ρίτσοντ. Εγώ είμαι εδώ από πλευρά του επόπτη προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων. Είμαστε ένα μικρό τμήμα των ενεχομένων σε αυτή τη διαδικασία. Συμβουλεύουμε για θέματα νομοθεσίας ε, σε διάφορους τομείς και είναι σαφές ότι και για τα νομοθετήματα προστασίας δεδομένων ε, δίνουμε τη γνώμη μας, είναι το βασικό μας καθήκον, γιατί εμείς επιτηρούμε και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Πολύ σημαντική είναι λοιπόν για μας όλη αυτή η συζήτηση, αλλά και γενικότερα. Οι συζητήσεις λοιπόν για τον νέο κανονισμό και τη νέα οδηγία. Νέος κανονισμός, νέα οδηγία. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία για την ε, συνεργασία των δικαστηρίων και των αστυνομικών αρχών. Στον τομέα. Αυτό βέβαια η επεξεργασία των δεδομένων είναι ε, ιδιαίτερα λεπτό θέμα. Καταλαβαίνετε όταν μιλάμε για αστυνομία. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν αυστηροί κανόνες προστασίας των δεδομένων για την αστυνομία. Αλλά βέβαια η αστυνομία πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει τις έρευνές της, να κάνει τη δουλειά της σωστά. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι υπάρχει και αυτή η πτυχή. Γενικά, πρώτον, να επανέλθω στη φύση του κειμένου, του κανονισμού. Μετά θα πω κάτι για το πεδίο εφαρμογής. Μετά θα μιλήσω για τα δικαιώματα των ε, υποκειμένων, των ατόμων δηλαδή. Μετά θα αναφερθώ στην ευθύνη των ε, οργανισμών που επεξεργάζονται τα δεδομένα, που είναι υπεύθυνα για τις βάσεις δεδομένων και μετά θα μιλήσω και για το σύστημα εφαρμογής από τις εθνικές και ενωσιακές αρχές, τις ανεξάρτητες αρχές λοιπόν προστασίας των δεδομένων. Αυτές οι ανεξάρτητες αρχές δεν υπάρχουν τόσο πολύ σε άλλους τομείς κοινωνικής δραστηριότητας. Και εδώ θα αλλάξουν πολλά στον τρόπο εφαρμογής. Πρώτον λοιπόν, ο κανονισμός. Η βασική αντίληψη της Αντιπροέδρου Ρέντινγκ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος νόμος σε όλη την Ένωση. Αυτό θα βοηθούσε και τις μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο που δεν τις απασχολούν λοιπόν τα εθνικά σύνορα. Ένας κανονισμός βέβαια σημαίνει ότι όπως λειτουργεί τώρα το σύστημα επιτρέπει κάποια ευελιξία στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν ε, τους ε, δικούς τους ε, κανόνες, τους δικούς τους κανόνες αλλά ούτως ώστε για παράδειγμα οι δημόσιες αρχές τους να έχουν κάποιους δικούς τους εθνικούς κανόνες είναι ε, ε, η τομή εδώ αρκετά λεπτή. Αλλά στόχος μας είναι να υπάρχει ένας κανονισμός για όλη την Ένωση. Ένας νόμος, αλλά θα υπάρχει κάποιο περιθώριο ελιγμών και στον ε, τομέα της υγείας και άλλους ευαίσθητους τομείς, απασχόληση για παράδειγμα. Πεδίο εφαρμογής. Ε, ξέρετε, είναι τόσο μακροσκελής ο κανονισμός, ε, 88 άρθρα, θα μπορούσα να μιλάω ώρες, αλλά θα επιχειρήσω να είμαι σύντομος. Πεδίο εφαρμογής. Η πρόταση της Επιτροπής θέλει να συμπεριληφθούν και οι μεγάλες εταιρείες στο ίντερνετ όπως το Google, το Facebook που δεν έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη. Συχνά την έδρα τους την έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει και αυτοί να συμμορφούνται προς αυτό το νόμο. Λέγεται λοιπόν στο νόμο ότι όσοι προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες της Ένωσης είναι επίσης υποκείμενα αυτού του κανονισμού. Πολύ σημαντικό αυτό. Αλλιώς η προστασία στο ίντερνετ θα ήταν ε, ιδιαίτερα ασαφής. Όπως υπόθηκε, ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνεται, αλλά η συνεργασία των αστυνομικών και δικαστικών αρχών όχι. Γιατί τώρα μπορούμε να το συζητήσουμε ώρες, αλλά εμείς ως επόπτες προστασίας δεδομένων θεωρούμε ότι δεν είναι η ιδανική λύση. Το λέμε καιρό τώρα. Αλλά αυτή η ε, θα πρέπει να τη δεχτούμε και να την εφαρμόσουμε στην εργασία μας. Είναι και θέμα βέβαια εκχώρηση κυριαρχίας τα θέματα αυτά αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Αυτό είναι πολύ λεπτό για τα κράτη-μέλη, γι' αυτό επελέγει αυτή η επιλογή που έχει τα θετικά τη. Τι διαπιστώνουμε τώρα. Διάφορες ομάδες πίεσης και ακόμη διάφοροι και εντός του Κοινοβουλίου θέλουν να εξαιρεθούν και κάποιοι άλλοι τομεί από το πεδίο εφαρμογή. Για παράδειγμα, ο χρηματοπιστωτικό τομέα επιχειρήθηκε να εξαιρεθεί είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι η προστασία των δεδομένων πρέπει να ισχύει για όλους τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας. Γιατί για όλους τους τομείς υπάρχουν κίνδυνοι σημαντικοί και παρόμοιοι. Γι' αυτό δεν θέλουμε να εξαιρεθούν άλλοι τομείς. Άλλο θέμα που έχει συζητηθεί πολύ εάν και κατά πόσο, η Ένωση ίδια θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στον κανονισμό. Διότι σε αυτή τη φάση εξαιρείται, δηλαδή η δραστηριότητα των θεσμικών οργάνων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η Επιτροπή δεν θέλει και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να υφίστανται τους ίδιους, να υπακούν στους ίδιους κανόνες. Αλλά είναι μακροπρόθεσμος στόχος να επιτευχθεί και για τη δραστηριότητα της Ένωσης το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Ακόμη, ο ορισμός των προσωπικών δεδομένων. Τι είναι προσωπικό δεδομένο. Και εδώ έχουν γίνει ατελείωτες συζητήσεις τα τελευταία 15-18 χρόνια. Τι αποτελεί προσωπικό δεδομένο. Ένα δεδομένο είναι προσωπικό μόνο όταν αναφέρεται ένα όνομα ή και αν έμεσα μπορεί να καθοριστεί ε, ποιο είναι, ποιος είναι, ποιο είναι το άτομο στο οποίο αναφέρονται κάποια στοιχεία. Θα πρέπει και αυτό να είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτό. Για παράδειγμα, γίνονται προσπάθειες από κάποιες ε, εταιρείε στο ίντερνετ να έχουν στοιχεία με κάποιο ψευδόνυμο. Και αυτά να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής. Αν δεν χρησιμοποιείς το δικό σου όνομα, αν έχεις ψευδόνυμο, θα πρέπει να έχεις την ίδια προστασία. Θέλουμε και προσπαθούμε να το επιβάλλουμε. Για τα δικαιώματα των υποκειμένων, προστασίες δεδομένων, όπως είπε και ο Ρίτσαρντ, είναι συνέχιση και βελτίωση της ήδη υφιστάμενης προστασίας. Εδώ, σε ένα σημείο όμως που υπάρχει σημαντική αλλαγή, είναι οι ευθύνε αυτών στις εταιρείες που επεξεργάζονται τα στοιχεία, που έχουν τις βάσεις δεδομένων, που ανταλλάσσουν στοιχεία. Εδώ υπάρχει μια μετατόπιση από κανόνες επιβολής σε ένα πιο γενικό σύστημα λογοδοσίας. Αφήνουμε περισσότερη ελευθερία δηλαδή στις εταιρείε σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουν τα δεδομένα, γιατί όλες οι εταιρείε δεν είναι ίδιες και η προστασία δεδομένων πρέπει να ισχύει και για τις μικρές εταιρείες και για τις τεράστιες εταιρείες στο ίντερνετ. Πρέπει να υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο θα συμμορφώνονται προς τον νόμο. Ένα άλλο σημαντικό θέμα συζήτησης. Από αυτούς τους ε, κανόνες που πρέπει να επιβάλλονται πρέπει να περάσουμε σε μια προσέγγιση που να βασίζεται περισσότερο στην εκτίμηση του κινδύνου και εδώ γίνεται συζήτηση. Αν περάσουμε σε μεθόδους εκτίμησης του κινδύνου, πώς ακριβώς θα, ε, ε, θα εξακριβώσουμε πώς εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες. Μεγάλη συζήτηση και αυτή. Μετά λοιπόν ε, τον επεξεργαστή, το υποκείμενο, το άτομο του οποίου είναι τα δεδομένα είναι το τρίτο ε, σημαντικό στοιχείο της νομοθεσίας. Πρέπει λοιπόν να συνδέεται η προστασία των δεδομένων του με τα βασικά δεδομένα, με τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματά του που προβλέπονται από την Ένωση. Άρα πρέπει ε, να υπάρχουν νόμοι και υπάρχει και νομολογία του ε, δικαστηρίου που καθορίζουν και το λέει και ο κανονισμός που προτείνουμε ότι οι οργανισμοί προστασίας των δεδομένων πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητοι από τους οργανισμούς και τους φορείς τους οποίους επιτηρούν. Η ανεξαρτησία λοιπόν των ε, φορέων προστασίας των δεδομένων είναι θεμελιώδες στοιχείο. Πρέπει να είναι οι φορείς αυτοί ανεξάρτητοι από εξωτερική ε, επιρροή, για παράδειγμα, πολιτικών οργάνων, για να έχουν δυνατότητα να επιτηρούν και να είναι απόλυτα εμπειρογνώμονες. τι θεωρούμε ότι το σύστημα της επιτήρησης μέσω των δικαστηρίων δεν λειτουργεί πάντα αποτελεσματικά γιατί είναι ιδιαίτερα λεπτό, ιδιαίτερα τεχνικό και λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το ίντερνετ ε, και η βάση δεδομένων, όλα αυτά δεν είναι ε, πάντα κατανοητά, χρειάζεται υψηλό επίπεδο γνώσης. Παραδοσιακά μέχρι τώρα και καταρχήν δεν θα αλλάξει αυτό. Η εποπτεία αυτή με βάση τους ενωσιακούς νόμους επαφίεται στους εθνικούς ελεκτικούς και ρυθμιστικούς φορείς. Αλλά οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς μέχρι τώρα είχαν απόλυτη ελευθερία δράσης και πολλές φορές για παρόμοιες περιπτώσεις κατέληγαν σε αντίθετα συμπεράσματα όπως για παράδειγμα για το Google Street View κάποιοι εθνικοί ρυθμιστές την επέτρεψαν αυτή την εφαρμογή και άλλοι όχι αυτή η κατάσταση λοιπόν δεν είναι ικανοποιητική. Το σύστημα λοιπόν τώρα προβλέπει μηχανισμούς για στενή συνεργασία των ε, ρυθμιστικών αρχών όταν τα θέματα αφορούν διάφορες χώρες, πολίτες από διάφορες χώρες. Και αν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ μερικών ε, ρυθμιστικών αρχών, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που να εγγυάται την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων. Καινοτομία λοιπόν του κανονισμού είναι ο, φορέας, ο Ευρωπαϊκός Φορέας Προστασία Δεδομένων που προτείνουμε που θα αντικαταστήσει την ομάδα εργασίας 29 είναι η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 αν δεν ξέρετε τι είναι είναι ένα δίκτυο αυτή η ομάδα εργασίας ε, των αρχών προστασίας των δεδομένων. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα σε ένα φορέα που θα μπορεί να δίνει τελειωτικές συμβουλές και ενδεχόμενα δεσμευτικές ή σχεδόν δεσμευτικές. Θα είναι λοιπόν ε, ρωμαλαίες γνωμοδοτήσεις για διάφορες δραστηριότητες των μεγάλων εταιριών ίντερνετ και θα μπορούν να πούν εάν είναι νομότυπες οι ε, δραστηριότητες αυτών των ε, οργανισμών και θα είναι εφαρμόσιμες οι γνωμοδοτήσεις τους για ολόκληρη την Ευρώπη. Να λοιπόν μια μεγάλη αλλαγή του νέου συστήματος. Αυτός ο φορέας δεν θα αντικαταστήσει τις εθνικές αρχές, αλλά θα χρειάζεται να συνεργάζονται στενά και να καταλήγουν σε λύσεις. Η εφαρμογή λοιπόν θα είναι πολύ πιο ρωμαλαία γιατί οι μηχανισμοί κυρώσεων θα ενισχυθούν ιδιαίτερα. Το ανέφερε ήδη ο Ρίτσαρντ σε, σε κάποια κράτη-μέλη. Οι δυνατότητε επιβολής ε, κυρώσεων των αρχών προστασίας δεδομένων είναι ανεπαρκής. Ο κανονισμός λοιπόν εναρμονίζει και ενισχύει το μηχανισμό επιβολής κυρώσεων Δεν θα μαλώνουν λοιπόν απλώς οι αρχές αυτές, θα δαγκώνουν. Και θα πονάει η δαγκωματιά. Γιατί προβλέπονται τρομερά πρόστιμα. Τρομερά πρόστιμα. Πολύ αποτελεσματικά. Γιατί ο κοινός μας στόχος είναι η εφαρμογή της προστασίας των δεδομένων. Αλλά ποιος είναι ο κύριος στόχος μας. Οι πολίτες μας. Εσείς, εγώ, όλοι μας να προστατευόμεθα επαρκώς όταν είμαστε στο ίντερνετ, όταν επεξεργάζονται κάποιοι τα στοιχεία μας, είτε είναι το μέσο της υγείας, τα στοιχεία μας, ε, τα υγειονομικά μας στοιχεία, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς, να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης και ενδεχομένων λαθών. Αυτό θέλει λοιπόν να κάνει η Κομισιόν. Οι συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ελπίζουμε να διατηρήσουν αυτόν τον ισχυρό μηχανισμό που προτείνεται. Ως επόπτες προστασίας δεδομένων θέλουμε να ενισχύσουμε τους κανόνες ούτως ώστε μέσω της νομοθετικής διαδικασίας να καταλήξουμε σε μια αρκετά ισχυρή πρόταση να μην αποδυναμωθεί η πρόταση που υπέβαλε η Κομισιόν. Ούτως έχουν τα πράγματα και με χαρά να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Έχετε παρακαλώ ερωτήσεις. Παρακαλώ σηκώστε το χέρι σας. Παρακαλώ. Στέφαν Όλιβ, είμαι ε, ελεύθερος επαγγελματίας, ρεπόρτερ για, από τις σκανδιναμικές χώρες. Η ελευθερία έκφρασης είναι το ερώτημά μου. Στο άρθρο 80, να με, να Στο άρθρο 80 αναφέρεται ότι ο κανονισμός δεν θα εφαρμοστεί για δημοσιογραφικές, καλλιτεχνικές και λογοτεχνικές δραστηριότητες ο επόπτης προστασίας δεδομένων τόνισε ότι δεν έχει έννοια στο σημερινό κόσμο γιατί όλοι περίπου ε, είμαστε επόπτες δεδομένων όταν είμαστε στο ίντερνετ. Ξέρετε, χθες είχαμε ένα τείχο Twitter. Θα ήταν εξαίρεση, θα εξαιρείται από τον κανονισμό ή θα καλύπτεται ο τείχος με Twitter που είχαμε χθες για παράδειγμα εδώ. Σε ποιον απευθύνεται την ερώτησή σας, ρωτάει ο συντονιστής. Σε όποιον από τους δύο θέλει να απαντήσει. Ε, από σκανδιναβική πλευρά το ερώτημα αυτό είναι σημαντικό, έχει συζητηθεί πολύ γιατί στις χώρες αυτές ε, η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής δραστηριότητας. Όταν μιλάμε για Twitter, για blog, ε, για όλα αυτά τα νέα μέσα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε πλήρως να ισχύει και για αυτά τα μέσα αυτός ο κανονισμός. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι δυνατή η επεξεργασία δεδομένων. Ότι δηλαδή δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε δεδομένα στο Twitter. Κοιτάξτε, Πολύ καλή ερώτηση, αλλά η απάντηση είναι αρκετά περίπλοκη. Ιδιαίτερα περίπλοκη. Το Twitter, για παράδειγμα, εάν το χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άτομο, αυτομάτως πρέπει να εξαιρείται για δημοσιογραφικούς λόγους. Αυτά τα νέα μέσα, τα εξατομικευμένα μέσα, επιτρέπουν αρκετή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Είναι λοιπόν τομέας που πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω τη θέση μας. Και αυτό που γίνεται στο facebook δεν είναι και πολύ διαφορετικό. το Facebook θα μπορούσε να εξαιρεθεί όχι για δημοσιογραφικούς αλλά για λόγους ατομικούς, για ιδιωτικές δραστηριότητες. Είπαμε ότι αν έχετε ένα κλειστό περιβάλλον φίλων δεν εφαρμόζεται το κανονισμό στο Facebook. Αν όμως έχετε απεριόριστο αριθμό φίλων στο ίντερνετ, αν έχετε ανοιχτές ρυθμίσεις για το Facebook σας, για τον ε, λογαριασμό σας του Facebook, τότε θα έπρεπε να ισχύει. Πρέπει λοιπόν για το Twitter να πούμε ότι αυτομάτως εφαρμόζεται ο κανονισμός, γιατί το Twitter είναι αυτομάτως ανοιχτό σε όλους. Δεν μπορεί λοιπόν να καλυφθεί από την εξαίρεση για ε, την ιδιωτική δραστηριότητα του νοικοκυριού. Ο κύριος Σόστακ, Το βασικό άρθρο είναι το άρθρο 80 στο άρθρο 80 προβλέπονται εξαιρέσεις από το γενικό κανόνα. Περί αυτού πρόκειται στο άρθρο 80. Το άρθρο 80 λοιπόν λέει ότι η προστασία των δεδομένων δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Χωρίς περιορισμούς. Υπάρχουν και άλλα δικαιώματα. Η ελευθερία έκφρασης. Στόχος μας λοιπόν είναι να καθορίσουμε ε, το διαχωρισμό μεταξύ αυτών των δύο δικαιωμάτων. Για την ελευθερία έκφραση συγκεκριμένα τι λέμε, ότι οι εθνικές παραδόσεις είναι εξαιρετικά διαφορετικές. Και γι' αυτό λέμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν κανόνες που να συνδυάζουν την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας με την ελευθερία έκφρασης με τον τρόπο που θεωρούν πιο σκόπιμο. Γιατί ο συνδυασμό ε, των δύο δικαιωμάτων αυτών στη Γερμανία είναι πολύ διαφορετικό από το συνδυασμό στην Εστονία. Και δεν υπάρχει αρμοδιότητα τη Ένωση για να καθορίσει την ελευθερία τη έκφραση. Άρα δεν μπαίνουμε σε αυτά. Αντίθετα με αυτά που λέμε στην οδηγία του 95, εδώ ενισχύουμε την πλευρά τη ελευθερία έκφραση. Γιατί στην προηγούμενη οδηγία έλεγε ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να προβλέψουν εξαιρέσεις για την ελευθερία έκφραση. Τώρα, στο 6ο του κανονισμού λέμε ότι θα προβλέψουν. Έτσι λοιπόν θα απαντήσω. Πρώτον, ενισχύουμε τους κανόνες ελευθερίας έκφρασης και δεύτερον, επαφίεται στις εθνικές παραδόσεις. Η συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν, στην, ε, απάντηση στην ερώτησή σας εξαρτάται από εθνικούς κανόνες. Αν θα καλυφθεί κάτι συγκεκριμένο από την ελευθερία της έκφρασης ή όχι, είναι θέμα εθνικής νομοθεσίας γιατί είναι θέμα του πώς ερμηνεύεται το καθαρά δημοσιογραφικός σκοπός από την εθνική νομοθεσία. Θα ήθελα να συνεχίσω την προηγουμένη ιδέα. Έχουμε μόνο πέντε λεπτά βέβαια. Εσείς εκεί κάτω. Όχι, εκεί, εκεί. Λέγομαι Πάρη Μάνικ, είμαι δημοσιογράφος από τη Φιλανδία και έχω ένα ερώτημα προς την Κομισιόν, αν δεν απατώμε. Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής ε, και ποια θεωρούνται θεμητά συμφέροντα του επόπτη. Αν θέλω να μαζέψω προσωπικά δεδομένα πελατών, μπορώ να επικαλεστώ θεμητό συμφέρον, τι θα πει ο επόπτης πού βρίσκονται τα όρια. Ε, ο άλλος εκεί κάτω, λέγομαι Λόσον, είμαι από την Εσθονία, από ένα εσθονικό περιοδικό και έχω ένα ερώτημα για την Wikipedia. Διότι λένε ότι και για αυτήν ισχύει κάποια δημοσιογραφική εξαίρεση. Αφού ισχύουν δημοσιογραφικές εξαιρέσεις, γιατί να μην ισχύουν και για τις εγκυκλοπαίδειες. Θα αρχίσουμε να σβήνουμε δεδομένα που έχουν αναρτηθεί εκεί αν κάποιος το ζητήσει. Θα αφαιρούνται και από τη Wikipedia δηλαδή. <clears throat> Στη Γερμανία υπήρχε μια περίπτωση όπου γνωστοί εγκληματίες δολοφόνοι εκείνοι που σκότωσαν δηλαδή ένα γνωστό ηθοποιό, ζήτησαν να αφαιρεθούν τα ονόματά τους από το σχετικό άρθρο της βικιπεδίας που αφορούσε τον ηθοποιό. Για μένα αυτό ξεπερνάει πολύ τα θεμητά όρια και θα ήθελα να ρωτήσω τι ισχύει ως προς αυτή την νομοθεσία. Μία ακόμη ερώτηση. με Παχάνε και έχω ένα ερώτημα για τη συγκατάθεση. Κύριε Σώστακ, μιλήσατε για ρητή και σαφή συγκατάθεση. Μου φαίνεται συνώνυμα λίγο πολύ αυτά τα δύο. Ισχύει αυτό ή όχι. Η κατάθεση αυτή όταν λέμε ότι πρέπει να είναι σαφής μπορεί να είναι και υπονοούμενη ή αυτό αποκλείεται από την ίδιο τον όρο σαφής. Okay, so I'll, I'll, Ας αρχίσω με το πρώτο και το τρίτο ερώτημα μαζί γιατί συνδέονται. Αφορούν τι καθιστά νόμιμη μια συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων. Αν ένα κράτος ή μια εταιρεία θέλει να συλλέξει δεδομένα πρέπει να είναι θεμητός ο λόγος. Ας δούμε με τα παραδείγματα και με τα συμφραζόμενα η σχέση μεταξύ του θεμητού συμφέροντος και της συγκατάθεσης είναι θέμα βαθμού. Αν ο αγοραστής δεν βλάπτεται στα προσωπικά του συμφέροντα, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά οι αρχές θα κρίνουν πότε υπάρχει παραβίαση και πότε όχι, πότε είναι θεμητό και πότε όχι δηλαδή. Παράδειγμα. Στο θέμα των άμεσων αγορών και μάρκετινγκ. Εκεί δεν χρειάζεται ρητή συγκατάθεση. Το Google όμως αν συνδυάσει δεδομένα προσωπικά για να κάνει profiling και στοχευμένη διαφήμιση τότε έχει συμβεί οι εποπτικές αρχές να πούν ότι απαιτείται ρητή συγκατάθεση για να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει, είναι θέμα βαθμού δηλαδή, με μονομένη περίπτωση συνδυασμού. Η συζήτηση για το θεμητό συμφέρον βασίστηκε στην έννοια του τρίτου. Δηλαδή, η Κομισιόν λέει πρέπει να, μπορεί κανείς να λάβει υπόψη του τα θεμητά συμφέροντα του επόπτη, οποιοδήποτε. Οποιαδήποτε οντότητος δηλαδή που έχει και εφαρμόζει ορισμένους κανόνες. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να λάβει υπόψη της και τα θεμητά συμφέροντα ενός τρίτου, δηλαδή κάποιου που δεν εφαρμόζει, δεν υπόκειται σε κανόνες. Λέμε λοιπόν ότι τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν εφόσον τα έχει στα χέρια του κάποιος επόπτης και εκείνου τα θεμητά συμφέροντα παίρνουμε υπόψη. Γι' αυτό λέμε ενός επόπτη όχι του επόπτη. Για τη συγκατάθεση τώρα, εδώ θέσατε τον δάκτυλων επί του τύπου των ύλων, δηλαδή όταν λέμε ρητό δεν εννοούμε υπονοούμενο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου δεν χρειάζεται συγκατάθεση και λέμε όποτε χρειάζεται τότε πρέπει να είναι ρητή. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνει ο άνθρωπος στον οποίο ζητούν τη συγκατάθεση ποιος είναι ο στόχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι για κάθε δοσοληψία θα χρειάζεται συγκατάθεση. αλλά για συγκεκριμένους στόχους. Θα μπορούσε κανείς με ένα και μόνο κλικ, με μία συγκατάθεση να χρειάζονται να χρησιμοποιείται αυτή η συγκατάθεση πολλές διαδικασίες, αλλά πρέπει να είναι πραγματική, ρητή και σαφή η συγκατάθεση. Τώρα για τη Wikipedia. Δεν είμαι βέβαια ο ίδιος επόπτης και δεν μπορώ να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα, αλλά για μένα επανερχόμαστε στο δύσκολο θέμα του πεδίου εφαρμογής, τι συμπεριλαμβάνεται, τι αποκλείεται. Είπαμε για ελευθερία έκφρασης, υπάρχουν εξαιρέσεις. Πολλά στη Wikipedia αφορούν το θέμα της ελευθερίας έκφρασης. Όταν όμως πρόκειται για ιστορικά δεδομένα, όπως το παράδειγμα που δώσατε, δεν είναι θέμα ελευθερίας έκφρασης. Είπαμε για την ελευθερία της έκφρασης υπάρχει εξαίρεση, αλλά υπάρχει και εξαίρεση για ιστορικά δεδομένα στατιστικά και για λόγους στατιστικής πληροφόρησης. Είναι βέβαια στόχος της ίδιας της ύπαρξης της Wikipedia να μην μπορεί κανείς να ξαναγράψει την ιστορία και να αλλάξει τα δεδομένα, τα αντικειμενικά δεδομένα. Αλλά βέβαια δεν έχουμε ακόμη συγκεκριμένα εργαλεία για να δούμε για αυτή συγκεκριμένα την περίπτωση τι μπορούμε να κάνουμε. Να προσθέσω μερικά σε αυτά που είπε ο Ρίτσαρντ. Όταν μιλάμε για συγκατάθεση, νομίζω τα είπαμε όλα. Αλλά τα άλλα δύο θέματα, για τα άλλα δύο θέματα θα ήθελα να πω ότι η προστασία των δεδομένων δεν είναι απόλυτο δικαίωμα που απαγορεύει την επεξεργασία, οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αλλά μόνο την περίπτωση όπου αυτό βλάπτει κάποιους. Χρειάζεται εδώ κάποια εξισορρόπηση λοιπόν. Όταν μιλάμε για το θεμητό συμφέρον, αυτό είναι φυσικά το πιο ακαθόδες θέμα σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών. Είναι όμως και το τελευταίο, έχουμε άλλα πέντε κριτήρια και ό,τι δεν βασίζεται σε αυτά το ανάγουμε στο θεμητό συμφέρον. Σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία και τον προτινόμενο κανονισμό απαιτείται μια εξισορρόπηση μεταξύ της ανάγκης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένα θεμητά συμφέροντα με το συμφέρον του ανθρώπου του οποίου συλλέγουν τα στοιχεία. Αν δεν υπάρχουν άλλα κριτήρια, χρησιμοποιούμε το κριτήριο του θεμητού συμφέροντος, με στόχο πάντοτε όμως την εξισορρόπηση. Αυτό ισχύει και για τη Βικιπέδια. Σαφώς είναι σωστό ότι εξαιρείται με βάση την ελευθερία του λόγου, αλλά Το γεγονός ότι οποιοδήποτε μπορεί να βάλει εκεί πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα σημαίνει ότι πρέπει να προστατεύονται οι άνθρωποι των οποίων τα ονόματα αναφέρονται ίσως με λανθασμένο τρόπο σε κάποιο άρθρο της βικιπεδίας. Και αυτοί οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να διαμαρτυρηθούν και να πούν ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν τα ονόματά τους με τρόπο σωστό ή θεμητό και μπορεί να προσφύγουν σε κάποιον επόπτη. Μπορούν να ζητήσουν δηλαδή, να διαμαρτυρηθούν γιατί χρησιμοποιήθηκαν τα ονόματά τους. Και εδώ πάλι χρειάζεται εξισορρόπηση μεταξύ διαφορετικών συμφερόντων. Ορισμένες εξαιρέσεις είναι βέβαια σαφείς και έτσι μπορεί η Wikipedia να λειτουργεί κανονικά. Απ' την άλλη όμως χρειάζεται και προστασία των προσώπων των οποίων αναφέρονται με λανθασμένο ή αθέμητο τρόπο τα ονόματα. Είναι δύσκολο θέμα η εξισορρόπηση βέβαια. Και γι' αυτόν τον λόγο και οι εποπτικές αρχές είναι τόσο σημαντικές. Υπάρχουν βέβαια πολλές περιπτώσεις, οποίες δεν μπορούμε όλες να προβλέψουμε εκ των προτέρων. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας και μπορούμε να περάσουμε τώρα στον επόμενο γύρο.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

Dzień dobry. Good morning. Bonjour. Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι οι άλλοι ομιλητές ε, του γύρου μας εδώ θα έρθουν ε, όταν πρόκειται να μιλήσει ο καθένας. Πρέπει να αρχίσουμε λοιπόν. Έχουμε τον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή. Θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση, εισαγωγικά σχόλια και μετά θα περάσουμε απευθείας στη συζήτηση, τις ερωτήσεις. Παρακαλώ, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, είναι απόλυτο δικαίωμά σας να θέσετε ερωτήσεις στον εισηγητή και τους άλλους ευρωβουλευτές που είναι αρμόδιοι για την εξέταση του θέματος και μπορείτε να θέσετε όχι μόνο νομικά, τεχνικά ερωτήματα αλλά και πολιτικής φύσης ερωτήματα. Οπότε, να σας παρουσιάσω τον κύριο εισηγητή, κύριο Γιάνν Φίλιπ Άλμπρεχτ των Πρασίνων, των Γερμανών Πρασίνων, εξελέγει πρώτη φορά το 2009. Είναι μέλος της Επιτροπής Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της ειδική Επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα και το ξέπλυμα χρήματος. Και αναπληρωτής ε, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και αυτό νομίζω βοηθάει. Και εδώ είναι και ο κύριος Kirkhope. Δεν είναι πρώτη φορά που μας μιλάτε για τέτοια θέματα. Είναι Βρετανός συντηρητικός ευρωβουλευτής είναι εδώ από την πλευρά των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Είστε αντιπρόεδρος επίσης της Ειδικής Επιτροπής για το Οργανωμένο Έγκλημα, τη Διαφθορά και το Ξέπλυμα Χρήματος. Είστε μέλος της Επιτροπής Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και είναι η τρίτη θητεία κατά την οποία είστε παρόν. Κύριε Άλμπρεχτ, παρακαλώ, Παρουσιάστε μας πώς έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Λίγα εισαγωγικά σχόλια για την άποψή μου για αυτήν την μεταρρύθμιση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Θεωρώ ότι ο στόχος αυτής της μεταρρύθμισης καθορίστηκε από ένα ψήφισμα που σχεδόν ομόφωνα ενέκρινε το Κοινοβούλιο του 2011, όπου τονίσαμε ότι η οδηγία του 95, η οδηγία 146, πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί έχουν ε, περάσει 18 χρόνια, έχουμε την εμπειρία της εφαρμογής της, αλλά και λόγω των εξελίξεων έκτοτε που δεν είναι μόνο τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά είναι και η επέκταση του ίντερνετ και η παγκοσμιμοποίηση. Έχουμε εταιρείες από όλο τον κόσμο που έχουν την έδρα τους εντός και εκτός της Ένωσης και μέχρι στιγμής ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες επεξεργασίας δεδομένων. Βεβαίως ε, για τις εταιρείε που ε, στόχος της δραστηριότητάς τους είναι επεξεργασία δεδομένων δεν είναι τόσο σημαντικό που έχουν έδρα. αλλά τα 500 εκατομμύρια πολιτών της Ένωσης δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Αν είστε Σουηδός για παράδειγμα και έχετε ένα iPhone και πάρετε, ε, αγοράσετε μια εφαρμογή app, ένα app από την Amazon δηλαδή, και αγοράσετε κάτι από το Amazon και σερφάρετε στο Google στο iPhone σας μέσω ενός browser που σας έχει πουλήσει μια εταιρεία. Η επεξεργασία δεδομένων μέσω όλων αυτών των φορέων δεν γίνεται με βάση το Σουηδικό νόμο προστασίας δεδομένων. Διότι η κοινωνική έδρα της εταιρείας ε, καθορίζει την ε, προστασία δεδομένων και είναι πολύ διαφορετικά τα μέτρα για την επεξεργασία δεδομένων ανάλογα από χώρα όχι μόνο για τις εταιρείε που πρέπει να συμμορφούνται με 27 διαφορετικές νομοθεσίες αλλά κυρίως για τα υποκείμενα, για τους πολίτες, τους καταναλωτές. Υπόκεινται σε πολύ διαφορετικούς κανόνες προστασίας δεδομένων. Οι διαφορές αυτές εξακολουθούν να ισχύουν διότι ο κανονισμός, η οδηγία συγγνώμη, έχει εφαρμοστεί από 27 εθνικά νομοθετήματα. Άρα δεν εφαρμόζεται επαρκώς αυτή η οδηγία. Βεβαίω υπάρχουν λοιπόν κανόνε προστασία δεδομένων, αλλά εφαρμόζονται και ερμηνεύονται με πολύ διαφορετικό τρόπο και πολύ διαφορετικό επίπεδο αποτελεσματικότητας. Θεωρεί λοιπόν το Κοινοβούλιο ότι εντάξει έπαιξε το ρόλο της αυτή η οδηγία, δεν διαμαρτύρεται κανείς για το περιεχόμενο της οδηγίας, αλλά διαμαρτύρονται πολλοί για τις διαφορές στον τρόπο εφαρμογής αυτής της οδηγίας και για το επίπεδο ακριβώς εφαρμογής. Γι' αυτό θέλουμε και ζητάμε ενιαίους κανόνες για όλη την ενωσιακή αγορά όσον αφορά τους κανόνες επεξεργασίας δεδομένων με βάση τους κανόνες που έχουμε από το 95. θέλουμε καλύτερη εφαρμογή θέλουμε ομοιόμορφη εφαρμογή και κυρώσεις και αυτό πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο κανονισμού του 2012 αλλά παραμένουν αρκετά θέματα ανοιχτά τα ανέφερα στην έκθεσή μου σε πολλά σημεία χρειαζόμαστε αλλαγές και στις 4.500 τροπολογίες που υποβλήθηκαν αναφέρονται και άλλα θέματα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα ακόμη ανοιχτά αλλά όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να προκύψει κανονισμός θα ήταν προστιθέμενη αξία, προστιθέμενο όφελος και για τους πολίτες αλλά θα ήταν και ένα μεγάλο βήμα ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς θα δημιουργούσε ισότιμο ανταγωνισμό για όλες τις εταιρείες και θα είχε ωφέλη και σε άλλους τομείς. Το δημόσιο τομέα, για παράδειγμα, όπου θα πρέπει να ευνοήσουμε την ανταλλαγή δεδομένων, κάτι που θα γίνει αν έχουμε κοινό σύστημα και κοινέ προδιαγραφές. Ευχαριστώ και να απαντήσω στις ερωτήσεις. Σας κύριος Κύρκο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Άκουσα την παρουσίαση του Γιάννης και θα προσπαθήσω να μην πω τα ίδια. Είναι προφανώς πολύ σημαντικό το ότι τώρα κάνουμε την αναθεώρηση της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων που για πρώτη φορά υποβλήθηκε πριν από 15-18 χρόνια. Τότε το ίντερνετ ζούσε την παιδική του ηλικία και δεν υπήρχαν τόσο πολύ κυβερνοέγκλημα. Τώρα όμως υπάρχουν δύο δισεκατομμύρια χρήστες του ίντερνετ και πάνω από ένα δισεκατομμύριο smartphones κυκλοφορούν. Το 1993 νομίζω ότι το ίντερνετ ε, ήταν 1% των επικοινωνιών, σήμερα φτάνει το 97%. Προφανώς λοιπόν χρειάζονται σαφέστεροι κανόνες που πρέπει φυσικά να εξυπηρετούν και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Αυτά τα δύο πρέπει να εξισορροπήσουμε με τον σωστό μέτρο αναλογικότητας. Εδώ βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και οι δοσοληψίες πρέπει να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία. Γνωρίζουμε βέβαια τη σημασία του γεγονότος ότι δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να φέρουν υπερβολικό βάρος γραφειοκρατικό και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει οι κανόνες να απλοποιηθούν και να εφαρμόζονται αναλόγως. 273 τροπολογίες έχουν κατατεθεί στην πρόταση κανονισμού. Η ομάδα μου υποστήριξε πολλές από αυτές, υπέβαλε πολλές από αυτές και κάναμε πολλές συνεδριάσεις μεταξύ Σκιωδών και του εισηγητή κ. Άλμπρεκτ για να διορθώσουμε ή να βελτιώσουμε τη διατύπωση. Και θα σταματήσω εγώ εδώ τονίζοντας ότι για μένα το σημαντικότερο είναι ότι χρειάζεται ένα σύστημα που να αποδίδει δικαιοδοσίες στα διοικητικά συμβούλια στους επόπτες να έχει τη δυνατότητα επιβολής προστήμων και φυσικά χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες γνωστοποίησης και αίτηση για πληροφόρηση και συνένεση, συγκατάθεση πρέπει να είναι σαφείς και ρητές. Δεν πρέπει να είναι οι διαφημίσεις που προβάλλονται υπερβολικές. Θέλουμε να αποφύγουμε την ρητή συγκατάθεση ως μόνο τρόπο χορήγησης κάποιας συγκατάθεσης και θέλουμε να βοηθήσουμε τους επόπτες στη δουλειά τους γιατί Νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθούν μεν οι δικαιοδοσίε τους αλλά να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Είναι δύσκολο πράγμα η εξισορρόπηση. Δεν νομίζουμε ότι πρέπει να είναι αυτόματο δικαίωμα η προσφυγή σε κάθε περίπτωση. Οι ενωσιακές υπηρεσίες πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα και βέβαια πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς και οι επόπτες πώς ακριβώς χρησιμοποιείται η συλλογή των δεδομένων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των μικρομεσαίων αυτών επιχειρήσεων και μέσω του ίντερνετ και γι' αυτό η ομάδα μου πρότεινε από τις 250 να φτάσουν στις 500 οι εξαιρέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βάση το μέγεθός τους και όχι μόνο τον αριθμό των δεδομένων που χειρίζονται. Εδώ θέλουμε διαφάνεια. Ε, όπως καταλαβαίνετε υπήρξαν πάρα πολλές εμπορικές πιέσεις και από λόμπι και για να προσθέσω στο θέμα της ξεσορρόπησης και εκτός Ευρώπης εξετάζονται όλα αυτά με ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον κόσμο ως πιθανό υπόδειγμα για την προστασία των δεδομένων. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι παράδειγμα χώρας όπου ήδη υπάρχει υψηλή προστασία και προστασία των δεδομένων καθώς και συγκεκριμένα κατά των γιγάντων όπως το Google Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε εφαρμόσουμε δεν θα βασίζεται απλώς στην αρχή του Safe Harbor που υπάρχει ήδη ως συμφωνία μεταξύ ΙΠΑ ΕΕ και Ένωσης αλλά εμείς θέλουμε μια νομοθεσία που να μπορεί να μεταφερθεί διεθνώς. Άρα πρέπει να είναι λογική και αναλογική και να υπάρχει και αποδοχή της από τους ενδιαφερόμενους και τους καταναλωτές αλλά και τις επιχειρήσεις που χρειάζεται πολλές φορές να συλλέγουν και να διατηρούν δεδομένα. Μάλιστα, αναφέρεστε νομίζω σε ένα άρθρο που δημοσίευσε χθες η International Herald Tribune που συζητούσε ακριβώς τη συζητούμενη αυτή νομοθεσία της Ένωσης την οποία προσέχουν διεθνώς και στην Νότια Αφρική συγκεκριμένα που προετοιμάζει και αυτή κάποια σχετική νομοθεσία και βασίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο. Το ίδιο ισχύει και για το Κατάρ και το Ντουμπάι. Έγινε και η διάσκεψη του Βερολίνου πριν από μερικές μέρες όπου ένα τρίτο των συμμετεχόντων ήταν από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον. Η Σόφη Ιντφελντ. Σας την καλωσορίζουμε. Είστε σκιώδη εισηγήτρια για τους φιλελεύθερους. και μέλος της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών. Και από καιρό κάνετε αγώνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θέλετε να πείτε τίποτα εισαγωγικά πριν αρχίσουν οι ερωταπαντήσεις. Ναι, ευχαριστώ καταρχάς. Ζητώ συγγνώμη που ήρθα με καθυστέρηση γιατί καμιά φορά είναι δύσκολο να τηρήσει κανείς ακριβώς το χρονοδιαγραμμά του. Λοιπόν, δεν άκουσα τα προηγούμενα, αλλά για περιοριστώ σε λίγα. Πρώτον, πάντοτε υπενθυμίζω ότι μιλάμε συχνά για προστασία ιδιωτικής ζωής ή αλλά αυτό που θέλουμε να προστατεύσουμε στην ουσία είναι ανθρώπους, δεν είναι το ίδιο. Ακούγεται σαν κάτι προφανές, αλλά δεν είναι. Θέλουμε να προστατέψουμε ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μόνο για ασφαλή διατήρηση των δεδομένων, αλλά και θέμα σεβασμού ελευθερίας του λόγου κλπ. Αυτά όλα καλύπτονται από την έκφραση προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Δεύτερον, πολύ συχνά οι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θεωρούνται φραγμός στην ελεύθερη επιχείρηση και στην σωστή εφαρμογή του νόμου, ενώ νομίζω ότι πρόκειται για το αντίθετο. Αν, υπάρχει, υπάρχουν επαρκείς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και άρα πρόκειται για προϋπόθεση για την σωστή χρήση τους. Τρίτον, η συζήτηση τονίζει κυρίως τον προετοιμαζόμενο κανονισμό και οι περισσότερες πιέσεις από τα λόμπι αυτό αφορούσαν. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη φάση στη δέσμη αυτή που είναι η οδηγία που υποτίθεται ότι καλύπτει όλους τους τομείς που έχουν εξαιρεθεί ή που εξαιρούνται μάλλον από τον κανονισμό. Την επιβολή του νόμου και την ασφάλεια, αν και οι χώρες μέλη πιέζουν αυτή τη στιγμή όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να εξαιρεθούν από τον κανονισμό και να μπουν στην οδηγία. Νομίζω ότι τελικά θέλουν να καταργήσουν πλήρως και την οδηγία ώστε να μην υπάρχει κανένας κανόνας προστασίας δεδομένων από τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές. Οι αρχές επιβολής του νόμου συνήθως χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από άλλους, από επιχειρήσεις, από τις τηλεπικοινωνίες, από τους επιβάτες, από γενικά εμπορικές δοσοληψίες από τράπεζες, όχι από τις ίδιες αυτές τις αρχές, δηλαδή την αστυνομία και τα δικαστήρια, οι οποίες αρχές, τα δικαστήρια και η αστυνομία δεν συλλέγουν πια δικά τους δεδομένα, μαζεύουν δεδομένα άλλων. Εμπορικά δεδομένα που μετά χρησιμοποιούνται για λόγους επιβολής του νόμου. Ενώ θα έπρεπε να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για τους δύο τομείς. Έπειτα. η διεθνής πτυχή. Όλοι μας νομίζω, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, αναγνωρίζουμε τη δυσκολία που έχει η επιβολή μιας νομοθεσίας για συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον. Είναι πολύ δύσκολο να περιοριστούμε σε συγκεκριμένο περιβάλλον και αυτό δεν αφορά πολιτικές ιδεολογίες, είναι τεχνική πρόκληση που έχουμε. και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τι θα πούμε για τη διεθνή μεταφορά δεδομένων εκτός Ένωσης. Και οι στενότεροι σύμμαχοι και φίλοι μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να συλλέξουν προσωπικά δεδομένα από μας ιδιαίτερα για λόγους επιβολής νόμου, αλλά καμιά φορά έχω το αίσθημα ότι όπως είδαμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες, ακόμη και απλοί πολίτες στις Ηνωμένε Πολιτείες έχουν αρχίσει να κουράζονται από την επιμονή αυτή των αρχών τους για τη συλλογή προσωπικών στοιχείων. Επίσης η διεθνής διάσταση είναι σημαντική και σε σχέση με κάτι που συζητάμε παράλληλα, δηλαδή την διατλαντική εμπορική, τις διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες που είναι κάτι το θετικό αλλά όπου πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η εμπορική αυτή συμφωνία δεν θα χρησιμοποιηθεί σαν νομικό τέχνασμα ή υπόβαθρο για να καλυφθούν απλά εμπορικά συμφέροντα χωρίς προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης πρέπει να επιλύσουμε τις διαφορές μας με τους Αμερικανούς ως προς το θέμα της πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρούνται στο Ευρωπα... στην Ευρώπη. Όχι στη ΣΥΠΑ, αλλά εδώ. Την πρόσβαση των Αμερικανών σε αυτά. Δηλαδή. Τέλος, ελπίζω οι κανόνες που θα εγκρίνουμε να μην αποτελέσουν φραγμό, αλλά μια πρόσθετη όθηση για την Ευρώπη, ώστε να προωθηθεί η οικονομία γενικότερα. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε παρακαλώ να πάρει πρώτος το λόγο. Και παρακαλώ όταν ε, θα πάρετε το λόγο να αναφέρετε το όνομα και το μέσο για το οποίο εργάζεστε. Παρακαλώ. Ε, και αν έχετε ερωτήσεις και από χθε ή από ε, νωρίτερα σήμερα το πρωί, παρακαλώ. Στέφαν Όλη, ανεξάρτητος δημοσιογράφος για τα σκανδιναβικά μέσα. Ο κανονισμός αυτός θα περιορίσει κάποιες προσβάσεις που έχουμε σε κάποιες χώρες σε επίσημα έγγραφα, κυβερνητικά site κτλ. Ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από αυτού, ξέρω ότι υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανονισμό. Θεωρείτε ότι αυτή η πλευρά του κανονισμού έχει κλείσει στην πορεία συζήτηση του κανονισμού ή μπορεί να αλλάξει. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ο κανονισμός προσπαθεί να, να προστατεύσει τα δεδομένα. Δεν είναι κανονισμός πρόσβασης στα έγγραφα Έχουμε άλλο κανονισμό για αυτό που έχει αναθεωρηθεί, υπάρχει και εθνική νομοθεσία. Άρα θα πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Η δική μου ερμηνεία για τις απόψεις που κυκλοφορούν είναι ότι κανείς δεν θέλει να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση σε έγγραφα με αυτό τον κανονισμό και αν έχει τέτοιο αποτέλεσμα ο κανονισμός που προτείνει η Κομισιόν θα τον τροποποιήσουμε για να διευκρινιστεί ότι θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα έγγραφα και μάλιστα θα πρέπει να βελτιωθεί. Είναι σαφές ότι η πρόσβαση σε έγγραφα πρέπει να υπόκειται σε κανόνες προστασίας δεδομένων. Αλλά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η προστασία δεδομένων για να απαγορευτεί η πρόσβαση στα έγγραφα, αλλά θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια την διαγραφή κάποιων προσωπικών δεδομένων πριν υπάρξει πρόσβαση σε κάποιο έγγραφο. Μπορούν να συνδυαστούν θαυμάσια οι προβλέψεις για αυτά τα δύο θέματα. Και φυσικά θέλουμε να τα συνδυάσουμε. Οι κανόνες προστασίας δεδομένων απλώς λένε ότι τα άτομα έχουν δικαίωμα προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Αλλά αυτό δεν πρέπει να παρεμποδίζει την πρόσβαση σε έγγραφα. Δεν την περιορίζει. Δεν θα περιοριστεί λοιπόν η πρόσβαση σε έγγραφα, αλλά είναι σαφές ότι αν θέλετε ένα έγγραφο για παράδειγμα για μια απόφαση δικαστηρίου πρέπει να προστατευτούν ε, οι παθόντες ή και οι μάρτυρες. Εάν λοιπόν δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον να του, δεν είναι προς το συμφέρον για παράδειγμα να είναι γνωστή η διεύθυνση κάποιων ατόμων που αναφέρονται σε ένα δικαστικό έγγραφο θα απαλληφθούν. Βέβαια, ο νόμος και τελικά τα δικαστήρια θα λύσουν το θέμα αυτό. Το Κοινοβούλιο δεν θέλει να περιορίσει την πρόσβαση στα έγγραφα. Τα προβλήματα αυτά υπάρχουν και με την ισχύουσα νομοθεσία θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Να προσθέσω, λέει ο κύριος Κέρχοπ, Πολλές χώρες της Ένωσης έχουν νόμους για την ε, ε, ελευθερία της πρόσβασης στην πληροφόρηση, πολύ εκτεταμένη ελευθερία πρόσβασης στην πληροφόρηση, αλλά υπάρχουν ε, και εθνικές αποφάσεις για αυτά. Ξέρετε ότι με τον Μάικλ Κάσμαν από την Σοσιαλιστική Ομάδα εξετάζουμε το θέμα της πρόσβασης των ενωσιακών, στα ενωσιακά έγγραφα. Εγώ είμαι υπέρ της ευρύτερη δυνατής πρόσβασης ε, σε ενωσιακά έγγραφα και με έχει απογοητεύσει η άποψη της Κομισιόν, η προσπάθεια της Κομισιόν να εισαγάγει πολλές εξαιρεσει σε αυτή την πρόσβαση. Θέλουμε τη μέγιστη διαφάνεια. Δεν θεωρώ ότι οι προτάσεις του Γιάνν, το κείμενο του κανονισμού, θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Κυρία Βέλ, συμφωνείτε? Συμφωνώ και με τους δύο ομιλητές δεν ε, εισάγουμε κενά δαιμόνια. Μπορεί να υπάρξει κάποια διαφορά μεταξύ του δικαιώματος στην προστασία του ιδιωτικού βίου και την πρόσβαση σε δεδομένα. Και υπάρχει και νομολογία για αυτά τα θέματα. Έχω αρκετή πείρα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κανονισμός για πρόσβαση έγγραφα και να σας πω ότι το πρόβλημα δεν είναι η νομοθεσία για, για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας, είναι η νοοτροπία των εθνικών κυβερνήσεων και της Κομισιόν. Υπάρχει μια κουλτούρα μυστικότητας. Εάν κάποιοι λοιπόν προσπαθούν να αξιοποιήσουν το νόμο για την προστασία δεδομένων για να μειώσουν την πρόσβαση έγγραφα, μα νοοτροπίας. Νίκλας Νίλσεν από το νέο παρατηρητή, New Observer. Ε, η ερώτησή μου είναι για την επιτήρηση μέσω του υπολογιστικού νέφους. Ε, ένας πρώην επικεφαλής ε, της υπηρεσίας μυστικότητας της Microsoft είπε ότι υπάρχουν πολλά κενά στο επίπεδο αυτό γιατί δεν αναφέρεται πουθενά στο κείμενο πρόβλεψη για το ασφαλή λιμένα. Μα δεν έχει να κάνει, λέει η κυρία Φαντβέλτ, ε, με τον ασφαλή λιμένα. Δεν, δεν δουλεύει αυτή η ιστορία του ασφαλή λιμένα. Πρόκειται για πλήρη σύγχυση. Στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε ένα νόμο που λέγεται ΦΑΙΖΑ. Ε, είναι ο, ε, η νομοθετική πράξη για την για, τα, για την ασφάλεια από εξωτερικές παρεμβάσεις έχουν νόμους που τους επιτρέπουν να σερφάρουν το υπολογιστικό νέφος και να ε, αξιοποιούν οποιαδήποτε στοιχεία οπουδήποτε. Οι δικές μας αρχές είναι ιδιαίτερα παθητικές. Ε, φυσικά είναι θέμα εξωταφικής εφαρμογής ε, νόμων των ΗΠΑ. Αλλά η Κομισιόν υπήρξε ιδιαίτερα απαθής και διαρωτώ τι θα κάνουν και οι κινέζικες αρχές. Θα ακολουθήσουν τόσο απαθή στάση ο κύριος Κέρκχοπ. Μα αναφέρθηκα στα θέματα του ασφαλούς λιμένα και προηγουμένως θέλω να πω ότι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ό,τι κάνουμε εδώ. Αναφερθήκατε μόλις στην Κίνα. Είναι πολύ σημαντικό ό,τι κάνουμε να διασφαλίζουμε ό,τι και κάνουμε σε ενωσιακό επίπεδο, να διασφαλίζουμε λοιπόν όσο γίνεται να εμπλέξουμε και άλλους. Πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο και οι αρχές των ΗΠΑ για οποιασδήποτε αλλαγές. Ήδη τους έχουμε συμβουλευτεί Πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια ούτω ώστε να είναι συμβατά αυτά που κάνουμε και με άλλους. Οι Κινέζοι οπωσδήποτε είναι ένας άλλος ε, σημαντικός παράγων. Εάν δεν τους ε, ε, εμπλέξουμε όλους, πολύ δύσκολο θα εφαρμοστεί διεθνώς οποιοδήποτε κανονισμός δικός μας. Ήρθε και ο κύριος Σον Κέλλιν. είναι συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής ε, Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κύριε Κέλλη, η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει. Ε, ίσως θα θέλατε να απαντήσετε και εσείς σε κάποιες ερωτήσεις που θα θέσουν δημοσιογράφοι. Έχετε άλλα σχόλια, άλλες ερωτήσεις. Θέλει κανείς άλλο το λόγο, παρακαλώ. Μίχαλ Μόσεκ, από το Τσεκ Daily πράβο. Χτες συζητήσαμε το θέμα της σχέσης της προστασίας των δεδομένων με τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος απάλληψης στοιχείων. Γιατί να μην πούμε απλώς ότι τα στοιχεία που εισαγάγει ο ίδιος ο χρήστης, για παράδειγμα, στο λογαριασμό του στο Facebook ή όταν ε, επισκέπτεται το Amazon, ή άλλα. Γιατί λοιπόν αυτά τα στοιχεία να μην είναι ιδιοκτησία του χρήστη που να αποφασίζει ο ίδιος πώς και σε τι βαθμό επιτρέπει τη χρήση τους και να έχει και το δικαίωμα να τα απαλείψει πλήρως. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Πρώτα απ' όλα να κάνω μια διευκρίνηση. Πολλές παρανοήσεις υπάρχουν γιατί δεν κατανοούμε όλοι πλήρως ε, όλα τα σημεία. Ορισμένα είναι σαφή. πολλοί κανόνες στην πρόταση κανονισμού. είναι και στον κανονισμό ή μάλλον στην οδηγία 46 του 95. Ισχύουν ήδη. Σε όλα τα κράτη-μέλη έχει εφαρμοστεί μέσω εθνικής νομοθεσίας αυτή η οδηγία. Άλλες χώρες καλύτερα, άλλες ε, χειρότερα, αλλά γενικά έχει εφαρμοστεί η οδηγία. Το δικαίωμα διαγραφής στοιχείων είναι τμήμα της οδηγίας στην ουσία. Ήδη υπάρχει και σε όλες τις εθνικές νομοθεσίες. Το δικαίωμα να ζητήσει κανείς διαγραφή όταν χορηγεί τα προσωπικά του στοιχεία σε κάποιον άλλον, λέγοντας ορίστε τα στοιχεία σας, μπορείτε να τα βάλετε στη βάση δεδομένων σας για να μου απαντήσετε για παράδειγμα. Και μετά μπορώ να ζητήσω τη διαγραφή τους. Εάν δεν υπάρχει λόγος να τα διατηρήσετε. Εάν δεν αναγκαίο να διατηρήσετε. Αυτό ισχύει ήδη στην νομοθεσία με πολύ λίγες εξαιρέσεις. Το θέμα που συζητάμε τώρα και είναι πολύ σημαντικό θέμα είναι τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν καταστεί δημόσια αν κάποιος ζητήσει την διαγραφή τους. Αυτό πρώτα απ' όλα είναι περίπλοκο τεχνικά, αν είναι ήδη σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, αλλά και λόγω άλλων ε, θεμάτων ελευθερία έκφρασης, ε, ελευθερία ενημέρωσης, του τύπου. Εισέρχονται εδώ και άλλα θέματα. Και είναι και πολύ ακριβό να γίνει κάτι τέτοιο, λόγω της τεχνικής φύσης. Αν κάποιος ζητήσει ήδη δημοσιευμένα στοιχεία να απαλληφθούν. Για παράδειγμα, εάν εγώ στείλω τα στοιχεία μου σε κάποιον και αυτός τα καταστήσει δημόσια χωρίς να με ρωτήσει και χωρίς να έχει νομικά θεμητό λόγο, οτιδήποτε γίνει παράνομα, φυσικά πρέπει μετά να διαγραφεί. Αυτό είναι κανόνας δικαίου που ήδη ισχύει με την τρέχουσα οδηγία. Το θέμα είναι αν εγώ ο ίδιος επιτρέψω την δημοσιοποίησή τους. Έχω μετά δικαίωμα να ξεχαστώ. Έχω δικαίωμα να τα διαγράψω. Και εδώ τίθεται το θέμα σε τι βαθμό Υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης για το δικαίωμα διαγραφής από τον ένα χρήστη στον άλλον. αν δεν καλύπτονται όλα αυτά από ε, κανόνες για ελευθερία έκφρασης, πρόσβαση σε έγγραφα κτλ. Θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Αυτό συζητάμε τώρα με αυτό το συμπληρωματικό δικαίωμα λύθης. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα, αλλά υπάρχει παρανόηση το δικαίωμα απάλληψης μη δημοσιοποιημένων στοιχείων ήδη υπάρχει και τηρείται. Κύριε Κέρκχοπ, γιατί πρέπει να φύγετε κατόπιν. Κέρκχοπ, να προσθέσω. Ο Γιάννα ανέφερε ήδη τους δύο σημαντικούς τομείς. Πρώτα απ' όλα το δικαίωμα λήθης. πρέπει να το ε, εξετάσουμε πολύ προσεκτικά γιατί μπορεί να έχει ε, επιπτώσεις ε, απρόσμενες πρώτα απ' όλα σε σχέση με τα κοινωνικά μέσα κάνουμε προτάσεις που να το κάνουν αυτό πιο εφαρμόσιμο αλλά και που τηρούν την αρχή της αναλογικότητας φυσικά πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις για λόγους δικαιοσύνης και αστυνομικών ερευνών κάθε είδους για θέματα ξέπλυματο χρημάτων, απατών κτλ. Βεβαίως καταρχήν κατανοώ αυτό το δικαίωμα αλλά πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις να προβλέπονται εξαιρέσεις που γενικά αναβασίζονται σε κοινή λογική. Το θέμα τώρα της συνένεσης και συγκατάθεσης είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Το 1995 είχε τεθεί το θέμα της χορήγησης αλλά δεν είχαμε τότε συμπεριλάβει τη λέξη ρητή συγκατάθεση. Τώρα την προβλέπουμε. Επειδή δεν είχε προβληθεί τότε είχαν υπάρξει ε, πολλές ε, και ε, δικαστικές υποθέσεις. Το εξετάσαμε προσεκτικά, ε, ζητήσαμε και τη γνώμη μόνον, Νομίζω λοιπόν ότι η συγκατάθεση πρέπει να έχει πολλές μορφές. Τις περισσότερες τις καλύπτει ήδη ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, πρέπει όμως να το επεκτείνουμε, ούτω ώστε η συγκατάθεση να μην είναι για όλα ρητή, εκπεφρασμένη, πρέπει να είναι κάπως ευρύτερο, να λάβει και άλλες μορφές. Είναι βεβαίως ιδιαίτερα λεπτό και περίπλοκο θέμα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ. Κυρία Ιντφελτ, μήπω θέλετε να Α, όχι, εσείς και ε, ε, κάτω. Να συνεχίσετε, ναι. Όχι, δεν ε, ρώτησα τίποτα για προσωπικά δεδομένα. Για, αλλά για όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προσωπικών δεδομένων. Γιατί, παραδείγματος χάρη, τι γράφουν συγκεκριμένα βιβλία όχι από άμεση συλλογή δηλαδή, αλλά από έμεση, από βιβλία μπορεί κανείς να δημιουργήσει προσωπικά δεδομένα. Τεχνικά δηλαδή δεν είναι προσωπικά δεδομένα, αλλά θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα προφίλ κάποιου από άλλες δημοσιεύσεις. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να φραγούν και αυτού του είδους τα δεδομένα. Κυρία παρακαλώ. Αυτό είναι, αφορά ακριβώς τον ορισμό των προσωπικών δεδομένων. Είναι μια άλλη από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό διακομματικά πάλι. Έχετε δίκιο. Είναι το θέμα αυτό της έμεσης συλλογής ή singling out. Η τεχνολογία επιτρέπει την ταύτιση ενός προσώπου με βάση στοιχεία που καθεαυτά είναι ανώνυμα ή τεχνικός ανώνυμα. Υπάρχει ένα γνωστό άρθρο πριν από δύο μήνες του Times της Νέας Υόρκης για ερευνητές που είχαν συλλέξει στοιχεία DNA ανώνυμα αλλά με μία απλή έρευνα στο Google μπορούσε κανείς να ταυτίσει τους κατόχους αυτών των στοιχείων DNA. Και χθες διάβασα πάλι κάτι. Φαίνεται ότι και απλώς και μόνο με τη βάση μηνυμάτων στον Twitter μπορεί κανείς να μαντέψει το φύλλο και την ηλικία αυτών που γράφουν τα μηνύματα. Και αυτό ήδη από τώρα. Άλλο τι άλλο ακόμη θα εμφανιστεί και θα εφευρεθεί. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτά που είπα πριν. Ίσως να μην πρέπει να μιλάμε για προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά προστασία των προσώπων. Πώς θα προστατευτούν οι άνθρωποι τα πρόσωπα κατά της αθέλητης αβούλητης χρησιμοποίησης των στοιχείων τους. Ο κύριος Σον Κέλλη. Πολύ σύντομο, ο κύριος Άλμπρεχτ μας είπε πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε και το δικαίωμα διαγραφής και λύθης είναι βέβαια απαράγραπτο. Η Κομισιόν πολλές φορές το έχει τονίσει και εκείνη, αλλά εξίσου σημαντικό θα ήταν να πούμε ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στα άκρα. Υπάρχουν και τα δικαιώματα της κοινωνίας γενικότερα ιδιαίτερα για τη διαγραφή ιδίω των εγκληματιών όσων έχουν ποινικό μητρό. Πρέπει να το εξισορροπήσουμε αυτό με την ανάγκη οι καταναλωτές να προστατευτούν, να διατηρηθούν τα δεδομένα για τους εγκληματίες, αλλά ο κύριος Άλμπρεχτ, για να μην δημιουργηθεί σύγχυση, προβλέπονται αυτές οι περιπτώσεις από τον κανονισμό εάν υπάρχει νομική υποχρέωση οποιαδήποτε χώρα να διατηρηθούν στοιχεία, τότε να υπάρχει σοβαρή νομική δικαιολόγηση. Αυτό λέει ο κανονισμός. Ακολουθώντας τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Άλλη παρεξήγηση. Για δημόσια αρχεία, για πρόσβαση σε έγγραφα, σε δημόσια έγγραφα, για τη λειτουργία δημοσίων αρχών, φορολογικών αρχών, αστυνομίας, οτιδήποτε, όλα αυτά θα διατηρηθούν όσο υπάρχει κατάλληλος νομικός λόγος, επαρκής νομικός λόγος. Αυτό ισχύει ήδη για όλες τις χώρες μέλη. Αυτό είναι σαφές όμως. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια βέβαια με βάση τα οποία Μπορεί να συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν στοιχεία αν υπάρχουν άλλα θεμητά συμφέροντα του επόπτη, αν υπάρχουν συμβόλαια κλπ. κλπ. Το δημόσιο συμφέρον δηλαδή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα. Αν εγώ ζητήσω διαγραφή ή δεν χορηγήσω τη συγκατάθεσή μου, πάλι μπορεί να πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα. Επομένως πρέπει να οριστεί ρητά, να οριστούν τα όρια της, του δικαιώματος στη διαγραφή. Αλλά η όλη συζήτηση φυσικά είναι λεπτό θέμα, ακόμη δεν το έχουμε πλήρως λύσει και υπάρχουν και ήδη όντως περιεχομένων ή πληροφόρηση που μπορεί να δημιουργήσουν προσωπικά δεδομένα από έμεσα στοιχεία. Αυτό ο επίσημος ορισμός όμως του προσωπικού δεδομένου είναι η βάση του κανονισμού. Οποιαδήποτε πληροφόρηση δεν καλύπτεται από τον ορισμό αυτό, δεν θα προστατεύεται. Και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο την πληροφόρηση περί προσώπων. Ορίστε εσείς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο Γιάννης Ρεζόπουλος από το Pathfinder στην Ελλάδα. Αν δεν είμαι ικανοποιημένος από τις εθνικές λύσεις για τα προσωπικά μου δεδομένα, έχω το δικαίωμα να προσφύγω στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ναι, έχετε. Γιατί πολιτικά είναι σαφές το θέμα. Υπάρχουν ορισμένοι που έχουν εκλεγεί από τους Ευρωπαίους πολίτες, εμείς δηλαδή οι εκπρόσωποι σας, και, πρέ... και οι εθνικοί βουλευτές και πρέπει να σας προστατεύουν καθώς και η κυβέρνησή σας. Νομικά αυτό επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, να μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη βασιζόμενη σε ένα ενιαίο νομικό εργαλείο σε όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή αγορά και αυτό θα ήταν μεγάλη πρόοδος και φυσικά θα αντικαταστήσει τους μεμονωμένους εθνικούς κανόνες που βασίζονται στην προηγούμενη οδηγία. Ο κύριος Κέλλη. Σωστό, σωστό. Αλλά θέλω να προσθέσω ότι ο όλος στόχος του κανονισμού είναι να υπάρξει ενιαίος, να υπάρξουν ενιαίοι κανόνες και στις 28 χώρες ενώ η οδηγία μπορούσε να εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο από την κάθε χώρα και μάλιστα και από ορισμένε περιφέρειες μέσα σε μια χώρα. Αυτή η μονοαπευθυντική θηρίδα One Stop Shop θα εφαρμόζεται ενιαία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν θα περιορίζεται σε εθνικούς κανόνες δηλαδή. και επομένως θα μπορείτε και να προσφύγετε. Σόφι Ινφελτ, μήπως θέλεις να προσθέσεις τίποτε στην ερώτηση του Έλληνα δημοσιογράφου. Μίλησα με τον Γιάννη εδώ συνεννοήθηκα και αν δεν είστε ικανοποιημένος από την απάντηση που θα σας δώσουν ο εθνικός σας επόπτης ή οποιοδήποτε άλλη εθνική αρχή, τότε μπορείτε να πάτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. ή σε άλλο εθνικό διαστήριο. Δεν θα υπάρξει όμως υπερεθνικός ενωσιακός επόπτης. Κοιτάξτε, γενικότερα και η Κομισιόν υποτίθεται ότι εκπροσωπεί το κοινό συμφέρον. Ναι, αλλά όταν βλέπω πώς προασπίστηκε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών γενικότερα η Κομισιόν, δεν θα στοιχημάτιζα ότι είναι και η αποτελεσματικότερη αρχή. Μάλιστα, άλλο ερώτημα. Η Σοφή Ιντφελντ μίλησε για το profiling από λογαριασμούς Twitter. Σημαντικό και αυτό. Πού βρίσκονται τα όρια μεταξύ των κοινωνικών μέσων και των υπολείπων μέσων. Τι θα καλύπτει και τι δεν θα καλύπτει ο κανονισμός. Το ρώτησα το ίδιο το πρωί και στην Κομισιόν και η απάντησή τους ήταν ασαφής. Πώς το ερμηνεύετε εσείς, κύριε Άλμπρεχτ. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή είναι η γκρίζα ζώνη ότι το εύρος, το πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού αφορά και τον ιδιωτικό οικογενειακό θα έλεγα τομέα αλλά μην εξετάζετε μόνο τον προτινόμενο κανονισμό αλλά και την ισχύουσα νομική νομοθεσία όπου σύμφωνα με την οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει εκδώσει αποφάσεις που λένε ότι οποτεδήποτε μπαίνει κάτι στο ίντερνετ πρέπει να γίνεται σεβαστός ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ακόμη και αν πρόκειται για μια μικρή κοινότητα 100 ατόμων, ό,τι μπαίνει σε μια ιστοσελίδα σημαίνει ότι είναι προσβάσιμο από πάρα πολλούς ανθρώπους. Με την ισχύουσα λοιπόν κατάσταση νομικά, όλα αυτά καλύπτονται από την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της οδηγίας του 95, όπως εφαρμόζεται εθνικά. Βέβαια τώρα το ξανασυζητάμε από την αρχή και από διαφορετική άποψη γιατί το ίντερνετ έχει πολύ πιο μαζικό χαρακτήρα από τότε. Και άρα δεν ίσως συμφωνούμε απόλυτα με αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσο και αν φύγεται αυτό από αυτή μας την άποψη. Γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια όρια, υπάρχουν προσδοκίες απρόσκοπτης πρόσβασης στο ίντερνετ. Αν βάλω κάτι στον Twitter, γιατί ήδη υπάρχει ένα θέμα προστασίας των μελών του Twitter. Αν βάλω κάτι λοιπόν στο Twitter και με, μου το διαβάσουν 300 άτομα, Πρόκειται ή δεν πρόκειται για γενική πρόσβαση. Είναι εμπορικό, δεν είναι εμπορικό. Όλα αυτά είναι ακόμη ασαφή, είναι η γκρίζα ζώνη. Πρέπει όμως να πούμε πολιτικά ότι μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου βάζουμε κάτι στο ίντερνετ όχι για όλους αλλά για συγκεκριμένες ομάδες, οικογένειες κλπ ε, τότε δεν θα καλύπτεται από τον κανονισμό. Αλλά δεν μπορούμε να το καθορίσουμε αριθμητικά. Αυτό θα το κάνει θέμα το θέμα με συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις το δικαστήριο. Είτε πρόκειται για φωτογραφίες γνωστών ανθρώπων όπως στις εφημερίδες. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε γενικά, αλλά περίπτωση με την περίπτωση. Η ερώτησή σας υπογραμμίζει την ανεπάρκεια του όρου επεξεργασία δεδομένων. Τι ακριβώς θέλουμε να προστατεύσουμε. Ό,τι βάζετε στο Twitter. Θέλετε να απαγορεύσετε την πρόσβαση ή τη χρήση των στοιχείων από κάποιον και για ποιο λόγο. Έχουν υπάρξει διάφορες ε, ε κατά του Twitter στις Ηνωμένε Πολιτείες γιατί η αστυνομία ήθελε πρόσβαση σε όλη την πληροφόρηση κάποιων λογαριασμών Twitter όχι μόνο το περιεχόμενο του ε, μηνύματος στο Twitter που ήταν βέβαια δημόσιο αλλά και την προσωπική πληροφόρηση, τα προσωπικά στοιχεία και έγινε μια συζήτηση και έχει ε, μάλιστα ε, αναφερθεί ο όρος η λογική προσδοκία προστασίας του ιδιωτικού βίου. Όταν βάζω κάτι στο Twitter θα ήθελα οι φίλοι μου ή και οι εχθροί μου γιατί έχω μερικούς ε, θα έπρεπε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία αλλά θα μπορούσε και η CIA να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία εναντίον μου. Ε, αυτά είναι θέματα που δεν έχουν ε, διευκρινιστεί. Ο κύριος Κέλλη, κυρία ε, Τβέλτ και εγώ σας παρακολουθώ. Κύριε Κέλλη, θέλετε να μας πείτε πώς βλέπετε αυτό το θέμα του Twitter, αλλά και γενικότερα να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για το Twitter. Είναι η δική σας απόφαση να βάλετε κάτι στο Twitter, δικό σας θέμα και θέλετε αυτοί που σας ακολουθούν, οι follower, να διαβάζουν αυτά που γράφετε και δεν είναι εύκολο μετά να ελέγξουμε τη χρήση αυτών των στοιχείων. Πρέπει λοιπόν να συζητηθεί το θέμα αυτό. Για τον ίδιο τον κανονισμό γενικότερα. Είμαι ο εισηγητής από πλευράς ε, της Επιτροπής Βιομηχανίας. και γι' αυτό ε, ήθελα να ρωτήσω τις επιχειρήσεις ποια είναι η άποψή τους και έκανα περίπου 250 συναντήσεις με διάφορες ε, ομάδες συμφερόντων από μεγάλες επιχειρήσεις, ε, μικρομεσαίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες καταναλωτών κτλ. Και καταλήξαμε σε μία πρόταση που πέρασε από την Επιτροπή μας και συζητώ τώρα με τον εισηγητή Γιάν Άλμπερτ στη συνέχεια της διαδικασίας. Ένας τομέας που με ανησυχεί είναι ότι ναι μεν έχουν καλές προθέσεις οι προτάσεις αυτές και είναι σκόπιμο να υπάρχει ομοιομορφία κανόνων στην Ευρώπη. Αυτό θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος τους, αλλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι το 99% των ευρωπαϊκών εταιριών, θα προκύψει κάποιο κόστος. Τώρα προηγουμένως είδα μια επισκόπηση του κόστους εφαρμογής των προτάσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου λέγεται ότι για όλες τις μικρομεσαίες το κόστος θα είναι κατά μέσο όρο 3.000 ευρώ για να συμμορφωθούν με τον κανονισμό. Να το έχουμε λοιπόν υπόψη μας αυτό όσο προχωράει η συζήτηση για να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ προστασίας των δεδομένων από τη μία αλλά προώθησης και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Γιατί ξέρετε είμαστε σε ύφεση, έχουμε απαράδεκτα υψηλή ανεργία στην Ένωση. Δεν πρόκειται οι υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν όλες αυτές τις θέσεις εργασίας που χρειαζόμαστε. Πρέπει λοιπόν για τις επιχειρήσεις που ξεκινάνε, για τα startup, να έχουμε συνέστηση ότι θα ε, υπάρξει κόστος για αυτές. Πρέπει να περιορίσουμε λοιπόν τις αρνητικές επιπτώσεις. Και βεβαίως να μην υπάρξουν και απρόσμενες επιπτώσεις. Βεβαίως όλες αυτές οι προτάσεις μπορεί να καταλήξουν ε, σε μια σωστή χρυσή τομή. Το βασικό είναι θέμα εμπιστοσύνης. Δεν πρόκειται να προκόψουν οι επιχειρήσεις εάν δεν τις εμπιστεύονται οι καταναλωτές. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ισχυρές οι ρυθμίσεις που προστατεύουν τους καταναλωτές χωρίς όμως να περιορίζουμε τις επιχειρήσεις. Δεν είναι σωστό. Και δεν νομίζω ότι είναι αντιφατικά αυτά τα δύο. Βεβαίω πρέπει να εμπιστεύονται οι καταναλωτές της επιχειρήσης. Αλλά και οι επιχειρήσεις μέσω της εμπιστοσύνη των καταναλωτών θα προκόψουν. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά είναι τα θέματα που με απασχολούν ως εισηγητή από πλευράς της Επιτροπής Βιομηχανίας. Ευχαριστώ. Έχουμε και την πλευρά των επιχειρήσεων λοιπόν και μάλιστα των μικρομεσαίων. Χαιρετίζουμε την παρουσία του κυρίου Δημητρίου Δρούτσα που είναι ο εισηγητής για την προστασία, για την οδηγία, για την προστασία των γενικών δεδομένων. Είναι μέλος ε, της σοσιαλιστικής ομάδας. Ήδη έχουμε εισέλθει στην ε, ουσία του θέματος Είστε αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και άρα και εσείς θα συμβάλλετε στη συζήτησή μας. Θα υπάρξουν τώρα ερωτήσεις και μετά μπορείτε και εσείς να παρουσιάσετε την άποψή σας. Η κυρία Τφέλντ. Έχετε κάτι να προσθέσετε. Αυτό που είπε ο Σον Κέλλη νομίζω είναι σημαντικό. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι τρομερή, είναι, <clears throat> αξίζει πολύ για τις επιχειρήσεις. Ας είμαι λίγο προκλητική. Ε, πολλοί αναφέρονται στο ενδεχόμενο κόστος για τις επιχειρήσεις αυτού του κανονισμού, αν να δούμε, και τα πιθανά κέρδη. Γιατί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι σίγουρα μεγάλο κέρδος. Κοιτάξτε, εάν οι επιχειρήσεις επρόκειτο να αποχωρούν από την Ένωση κάθε φορά που εγκρίνουμε κάποιο νομοθέτημα δεν θα μας είχαν μείνει καθόλου επιχειρήσεις. Κάθε φορά που μιλάμε για κοινωνικά δικαιώματα, κάθε φορά που μιλάμε για περιβαλλοντικά δικαιώματα, πάντα έρχονται και λένε «Ω, καταστροφή, θα σηκωθούμε να φύγουμε». Θα σηκωθούν να φύγουν από μια αγορά 500 εκατομμυρίων κατά μέσο όρο πολύ ευπόρων καταναλωτών. Αν ακούσετε τι έλεγαν οι επιχειρήσεις για τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, μας έλεγαν ότι θα καταστραφεί πλήρως η βιομηχανία, μας έλεγαν. Θα καταστραφούν πλήρω οι επιχειρήσεις μα. Μία γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει τεράστια κέρδη. Είχαν τα υψηλότερα κέρδη ανατρίμηνο της ιστορίας τους πρόσφατα. Μέσω της χρήσης των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ως κινήτρου για καινοτόμες για την εισαγωγή καινοτομιών στην ε, δραστηριότητά τους. Μπορούν να αξιοποιήσουν λοιπόν την νομοθεσία μας και με θετικό τρόπο. Και τέλος, πολύ συχνά οι κανονισμοί για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας ε, εμφανίζονται στην Ευρώπη σαν να είναι ιδιαίτερα ε, αυστηροί ενώ για παράδειγμα στις ΗΠΑ λέγεται ότι είναι πολύ χαλαροί. Δεν ισχύει αυτό. Εάν κάνουμε μια μελέτη συγκριτική θα δείτε ότι και στι ΗΠΑ υπάρχουν πολύ αυστηρέ προδιαγραφέ και συνέχεια περνάνε και νέα νομοθετήματα προστασία τη ιδιωτική σφαίρα. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο δικό μα επίπεδο προστασία των ιδιωτικών δεδομένων. Παρακαλώ, η Βασιλική. Ευχαριστώ. Βάλια Καϊμάκη από την ε, ελληνικό ραδιόφωνο, την ΕΡΑ. Έγιναν πολλές τροπολογίες στην αρχική πρόταση Επιτροπής. Θα ήθελα να μου συνοψίσετε αν υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία ή αν απλώς ε, έγιναν τεχνικές τροποποίησεις. Υπάρχει διαφορά αντίληψης μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Είναι τόσο έντονες διαφορές που οι δύο οδηγίες δεν θα μπορέσουν να ε, συνεπάρξουν. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Κοιτάξτε, να διορθώσω πρώτα απ' όλα. Είναι ένας κανονισμός και μία οδηγία. Ένας κανονισμός και μία οδηγία. Ναι, ε, μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Για την ερώτησή σας. Ο κανονισμός θίγει πολλές πλευρές ε, της ζωής μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι μόνο τεχνικό θέμα. Είναι πολιτικό θέμα, αφορά τη ζωή μας, αφορά όλους μας. Αφορά τους ανθρώπους, την κοινωνία, το πώς συνεπάρχουμε. Φυσικά προκύπτουν λοιπόν και πολλές ανησυχίες. Ορισμένες ε, τις έχει αντιμετωπίσει η πρόταση της Κομισιόν, αλλά δεν ξέρω εάν όλοι ε, τη διάβασαν πλήρως, ε, αν την κατανόησαν πλήρως, αν γνωρίζουν την ισχύουσα νομοθεσία Ήδη διευκρινίζουν αυτά τα υπάρχοντα κείμενα πολλά θέματα, αλλά υπάρχουν και θέματα που δεν τα έχει αντιμετωπίσει η πρόταση της Κομισιόν, αλλά δεν την έχουμε ακόμη εγκρίνει. Θα βελτιωθεί λοιπόν αυτή η πρόταση. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά κάποιες αναλυτικές ε, διατάξεις για ορισμένα θέματα που δεν μας έχουν απασχολήσει τόσο πολύ στο παρελθόν. Ο κόσμος μας, όπως ξέρετε, είναι διασυνδεδεμένος, παγκοσμιοποιημένος Έχουμε κράτη δικαίου, δημοκρατική οργάνωση των κοινωνιών μας και η επίλυση όλων των ε, ζητημάτων που προκύπτουν είναι δυσχερής. Αλλά μπορεί να γίνει. Καλή είναι η πρόταση της Επιτροπής, έχουν υποβληθεί μερικές καλές τροπολογίες που βελτιώνουν το κείμενο, αλλά όπως ξέρετε δεν ε, ξεκινάμε εκ του μηδενός. Το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό. Στο Κοινοβούλιο είχαμε και το ψήφισμα του 2011 που τονίζει τι θέλουμε να βελτιώσουμε. Η οδηγία 4695 δεν θα αντικατασταθεί από κάτι εντελώς διαφορετικό. Αντίθετα, είναι το σημείο εκκίνησής μας. Θέλουμε να τη βελτιώσουμε. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι το εντελώς διαφορετικό και καινούριο. Υπάρχει ε, συναντήληψη για τα θέματα αυτά στο Κοινοβούλιο. Στις επιμέρους διατάξεις βέβαια θα δούμε τι έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα, τι θέλουμε περαιτέρω να επιτύχουμε, νομίζω ότι θα καταφέρουμε ε, να καταλήξουμε στις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο γιατί έχουμε κοινέ ανησυχίες. Ελήφθησαν αποφάσεις με ευρύτατη πλειοψηφία που λένε ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο κανονισμό θα έχει και θετική οικονομική επίπτωση. Δεν θα υπάρξει μόνο κόστος, θα υπάρξει και τεράστιο όφελος από έναν ενιαίο κανονισμό θα ολοκληρώσει την ενιαία αγορά, θα προκαλέσει και οικονομική ανάπτυξη και καινοτομίε, θα αυξήσει την εμπιστοσύνη όχι μόνο και των καταναλωτών αλλά και των νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ξέρουν ότι εφόσον θα τηρούν τον κανονισμό δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Θέλω λοιπόν να καταλήξω με αυτήν την πολύ θετική και αισιόδοξη προοπτική θα επιτύχουμε συμβασμούς για να αντιμετωπιστούν όλες οι λογικές ανησυχίες πολλών πλευρών. Ήδη θεωρώ ότι θα καταλήξουμε σε σκόπιμες λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντρούτσα, σας παρακαλώ. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει και ελληνική διερμηνία. Ε. Uh, uh, Δεν διαφωνώ με τον Γιάννα Άλμπρεχτ. Πολύ καλά μας τα είπε. Όντως, συζητήσαμε πάρα πολύ μεταξύ μας. Θα επανέλθω αργότερα στο δεύτερο τμήμα της νομοθεσίας προς το παρόν για το συγκεκριμένο ερώτημα των διαφορετικών αντιμετωπίσεων στα τεχνικά τουλάχιστον θέματα. Εγώ είμαι κανονικά ο διπλωμάτης, πρέπει να θεωρούμε λόγω του παρελθόντος μου, αλλά ο Γιάννα Άλμπρεχτ υπήρξε πολύ διπλωματικότερο από αυτά που θα πω τώρα. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτές τις συζητήσεις και εδώ μέσα με τις τροπολογίες βλέπουμε κάτι πολύ καθαρά. Το όλο θέμα της μεταρρύθμισης της προστασίας των δεδομένων είναι πώς θα εξισορροπήσουμε την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών από τη μία και των συμφερόντων των επιχειρήσεων από την άλλη. Αυτό είναι το όλο θέμα. Προσωπικά από τις συζητήσεις εδώ και τόσους μήνες και από τις εκατοντάδες και χιλιάδες τροπολογίες βλέπω πως μερικές επιτροπές του Κοινοβουλίου ψήφισαν μέχρι τώρα και βλέπω, φοβάμαι ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα πράγματα. Βλέπω δυστυχώς μία κίνηση προς την προστασία των συμφερόντων των επιχειρήσεων κυρίως. Το ξαναλέω η πολιτική μου ομάδα, οι σοσιαλιστές δηλαδή, και εγώ προσωπικά δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι ή τουλάχιστον καθόλου ικανοποιημένοι με αυτή την τάση. Γιατί σε αυτό το θέμα της προστασίας των δεδομένων οι πολιτικές ιδεολογίες έχουν πια αποκρισταλωθεί. Σιγά σιγά βλέπουμε να δημιουργούνται κόκκινες γραμμές που δημιουργούν οι διάφορες πολιτικές ομάδες και εγώ διακρίνω μια αλλαγή προς μάλλον την προστασία των επιχειρήσεων παρά των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Για μένα λοιπόν είναι μια αλλαγή της Διοντολογίας της φιλοσοφίας ή της ιδεολογίας όπως θέλετε και όχι μόνο στο τεχνικό επίπεδο βέβαια υπάρχουν εκατοντάδες τροπολογιών και στο τεχνικό θέμα αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές πρόκειται και για μεγάλη ιδεολογική πολιτική διαφορά εσείς εκεί κάτω είχατε πει είχατε εκφράσει μια ανησυχία κατά πόσον η δέσμη θα εγκριθεί τώρα ή αν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολλά χρόνια ακόμη. Εγώ συμφωνώ με τον Γιάνν Άλμπρεχτ. Νομίζω ότι θα κατορθώσουμε να πετύχουμε τους απαραίτητους συμβιβασμούς για να εγκριθεί, αλλά φοβάμαι ότι μερικές χώρες μέλη στο Συμβούλιο μπορεί να μην τηρήσουν την ίδια στάση ή να μην ενδιαφέρονται τόσο πολύ να περάσει η δέσμη πριν τη λήξη αυτής της θητείας του Κοινοβουλίου. Θα φανεί βέβαια αυτό. Μόλις αρχίσει ο τριμερής διάλογος, ελπίζω να αρχίσει, θα δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις στο Συμβούλιο. Και τότε καθήκον και των πολιτών ως κοινή γνώμη θα είναι να εκφράσουν την άποψή τους και να ασκήσουν και την απαραίτητη πίεση στις κυβερνήσεις τους, σε ορισμένα κράτη-μέλη τουλάχιστον, που και θέλουν να κερδίσουν απλώς χρόνο για να καταλάβουν ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και δεν πρέπει να παίζουν παιχνίδια. Για το δεύτερο θέμα αργότερα. Κύριε Κέλλη για αυτή τη γενική προσέγγιση και την πολιτική αλλαγή που ανέφερε ο κύριος Δρούτσας, τη βλέπετε κι εσείς. Πρώτον, δουλειά της Κομισιόν είναι να προτείνει την ομοθεσία και του Κοινοβουλίου να την αναλύσει, να την εξετάσει, να την τροποποιήσει ή να την απορρίψει. Δεν νομίζω βέβαια ότι θα απορριφθεί γιατί οι περισσότεροι ανεξαρτήτως ιδεολογίας θεωρούν ότι ένας ενιαίος κανόνας για ολόκληρη την Ευρώπη είναι κάτι καλύτερο από 28 διαφορετικούς και αυτή η μονοαπευθυντική θηρίδα που είπα και πριν είναι κάτι θετικό για τους πολίτες. Γενικά λοιπόν οι περισσότεροι συμφωνούν τώρα στις λεπτομέρειες, εκεί υπάρχουν οι δυσκολίες. Βέβαια έχουμε διαφορές ως διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Άλλα φρονούν οι χριστιανοδημοκράτες, άλλα οι σοσιαλιστές, άλλα οι πράσινοι. Αλλά επίσης και μέσα στην κάθε ομάδα υπάρχουν διαφορές. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να συνδυαστούν και αυτή ακριβώς είναι η δουλειά του εισηγητή ο οποίος την φέρνει σε πέρας μέχρι τώρα πολύ ικανοποιητικά. Έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις μεταξύ σκιωδών, δεν μπορώ να τις συνοψίσω σε μια φράση, αλλά νομίζω ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία και θα προχωρήσουμε θα με απογοήτευε ιδιαίτερα, θα θεωρούσα μάλιστα ότι έχουμε σπαταλήσει δυόμιση χρόνια χωρίς κανένα λόγο, αν τελικά δεν γινόταν δεκτή η δέσμη. Και πρέπει να τελειώσει η ανάλυση σε αυτή τη θητεία. Η Ιρλανδική Προεδρία κάνει ό,τι μπορεί είναι από τις προτεραιότητες της το θέμα, γιατί αν περάσει το θέμα μέχρι την επόμενη θητεία μετά τις ευρωεκλογές, Νομίζω ότι θα ήταν αρνητικό για όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ιντφελτ, εσείς πώς το βλέπετε πολιτικά. Υπάρχει αλλαγή. Καταρχήν πριν απαντήσω σε αυτό θα ήθελα να επαναλάβω ότι πρέπει να διαλύσουμε αυτόν τον μύθο ότι είτε είμαστε υπέρ των ανθρώπων είτε υπέρ των επιχειρήσεων. Και αν είμαστε υπέρ των επιχειρήσεων αν είμαστε υπέρ των επιχειρήσεων, τότε αυτόματα είμαστε και υπέρ των καταναλωτών. Τι λέει ο κόσμος, ότι θέλει τα δεδομένα του να είναι ασφαλή. Αλλά να υπάρχει και προσφυγή σε περίπτωση παρανομίας. Δεν θα έπρεπε να τα βλέπουμε λοιπόν ως απόλυτα διαφορετικά θέματα. Έχουν μείνει λίγοι πια φιλελεύθεροι βέβαια γενικώ μετά τη δημοσιονομική κρίση, αλλά πρέπει όλες οι ομάδες αμοιβαία να ενισχύονται αφού συμφωνούν στα βασικά. Ο Κέλλη έχει δίκιο ότι η δέσμη θα περάσει, το θέμα όμως είναι με τι μορφή. Θα υπάρξει καμία ουσιαστική βελτίωση ως προς την υπάρχουσα κατάσταση, περιθωριακή βελτίωση ή υπαναχώρηση. Αυτό είναι το θέμα. Ελπίζω να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση γιατί η δέσμη ολόκληρη δεν είναι κάτι επαναστατικό και τελείως καινούριο που μόλις το σκεφτήκαμε. Βασίζεται στην υπάρχουσα νομοθεσία η οποία βέβαια πολλές φορές δεν εφαρμόζεται καθόλου ούτε από τις δημόσιες αρχές ούτε από τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό λέμε ότι δεν θέλουμε μόνο νομοθεσία προσαρμοσμένη στην εποχή μας, αλλά και πραγματική εφαρμογή της. Ας πούμε το δικαίωμα της διαγραφής. Ή τώρα το λέμε της λύθης. Αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Να δούμε ψυχρά με ψυχραιμία πώς έχουν τα πράγματα και τι προσδοκίες έχουν οι καταναλωτές και οι πολίτες από τις δημόσιες αρχές. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει οι κυβερνήσεις ιδίω να σκεφτούν πολύ καλά τα πράγματα πριν αποδυναμώσουν τις προτάσεις μας. Μήπως κύριε Άλμπρεχτ μου θέλετε να κάνετε κανένα σχόλιο για αυτό το πολιτικό θέμα. Εξάλλου, τι φρονείτε για το Συμβούλιο και την Ιρλανδική Προεδρία και το πώς χειρίζονται το θέμα. Ποια είναι η ισορροπία των δυνάμεων. Ξαναλέω σαφέστατα. Ευρύτατη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο υπήρξε για να τονιστεί ότι δεν θέτουμε ένα αμφιβόλο την οδηγία του 95 που ισχύει και έχει μεταγραφεί σε εθνικά νομοθετήματα. Αυτή είναι η βάση επί της οποίας οικοδομούμε. Δεν οπισθοδρομούμε. Και το είπε επανειλημμένα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κανένα κράτος δεν το αμφισβητεί. Άρα και το Συμβούλιο το έχει τονίσει. Έχουμε λοιπόν μια κοινή βάση. Να μην παραβλέψουμε ωστόσο ότι υπάρχουν πολλοί που θέλουν να υπάρξει οπισθοδρόμηση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Αν κάποιες επιχειρήσεις εκτός ένωσης δραστηριοποιούνται στην αγορά μας χωρίς να σέβονται την νομοθεσία μας, δεν θα ε, προσαρμόσουμε εμείς την νομοθεσία μας στη δραστηριότητά τους, αλλά αντίστροφα. Ενισχύουμε λοιπόν ακριβώς την νομοθεσία μας. Και εδώ εκνευρίζομαι, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι προτείνουμε συμπληρωματική γραφειοκρατία και κόστος. Όχι. Ως εισηγητής προσπαθώ να εναρμονίσω την υπάρχουσα νομοθεσία, ούτω ώστε να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή της εσωτερική αγορά. Αυτό κάνω. Τίποτα περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο. Δεν νομίζω ότι είναι παράλογα αυτά που κάνουμε, ούτε ασήμαντα, είναι και λογικά και σοβαρά. Όλοι πρέπει να το καταλάβουν παντού στον κόσμο και όλοι οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές πρέπει να ακολουθούν αυτή την προσέγγιση για την εργασία μας. Και όπως είπα, με ενοχλούν κάποιες τροπολογίες που απλώς αμφισβητούν αυτό που ήδη υπάρχει. Μα δεν θέλουμε να το αμφισβητήσουμε, θέλουμε να το ενισχύσουμε, να το βελτιώσουμε. Και επίσης ε, να αναπτύξουμε και νέους τομείς. Η, ε, ε, η θελημένη ιδιωτική, προστασία της ιδιωτικής σφαίρας, η εξορισμού προστασία της ιδιωτικής σφαίρας, το δικαίωμα στη λύθη, Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτό το δικαίωμα διαγραφής που ήδη υπάρχει δηλαδή. Να δούμε και τα όρια του όταν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία. Έχει κάποια όρια. Υπάρχει και θέμα ελευθερίας ε, έκφρασης. Αυτό περιορίζει το δικαίωμά μου ε, να ξεχαστώ. Τα έχουμε αυτά στην υπάρχουσα νομοθεσία. Την ίδια ερμηνεία θα υιοθετήσουμε Πιστεύω ότι υπάρχει πλειοψηφία και στα τρία βασικά όργανα υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών. Τουλάχιστον έτσι έχουν πει. Βέβαια, τίθεται το ερώτημα. Όντως το πράττουν κιόλα. Στοχεύουν σε ένα αποτέλεσμα που θα το επιτύχει. Όπως είπε και η κυρία Εντφέλντ, το αποτέλεσμα έρχεται στο τέλος. Δεν είμαι σίγουρος ότι και τα τρία θεσμικά όργανα ε, το επιδιώκουν. Ίσως υπάρχει κάποια ασάφεια. Γιατί πραγματικά διαρωτώ με τι είδους πολιτικά κόμματα, τι είδους, τι είδους πολιτικοί άνδρες και γυναίκες είναι αυτοί που ένα λένε και άλλο κάνουν. Δεν θέλουμε να θίξουμε την ψηφιακή αγορά, αλλά έχουμε ένα δημοκρατικό σύστημα, έχουμε πολιτικούς, έχουμε ηγέτες και όλοι θα πρέπει να σέβονται και να προασπίζουν τα δικαιώματα των πολιτών όπως και στα κράτη-μέλη. Και πρέπει να επιτύχουμε αυτό που περιέχει το ψήφισμα του 2011. Ορίστε σαφής και ιδιαίτερα πολιτική απάντηση στο βασικό φιλοσοφικό ερώτημα. Ο κύριος Ρούτσας. Συμφωνείτε? με αυτά που είπε ε, τα πολύ κατηγορηματικά ο προηγούμενος. Μα πάντα συμφωνώ με τον Γιάνν Άλμπρεχτ. Τα συζητήσαμε όλα αυτά ενδελεχέστατα. Έχουμε έναν αγωνισμό λοιπόν και μία οδηγία, αλλά ξέρετε ότι από την αρχή το Κοινοβούλιο ήθελε να υπάρξει ένα μέσο, ένας κανονισμός που να καλύπτει όλους ε, τους τομείς της προστασίας δεδομένων. Δυστυχώς η Κομισιόν επέλεξε άλλη μέθοδο κανονισμού και οδηγία για τον τομέα εφαρμογής του νόμου και αστυνόμευσης. Όπως έχω πει επανειλημμένα, δεν μας ικανοποιεί αυτή η λύση ως κοινοβούλιο, αλλά είμαι ρεαλιστής. Έχω διατελέσει και υπουργό Ξέρω τις ευαισθησίες ε, και τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου, οπότε η απόφαση της Κομισιόν να διαχωρίσει κανονισμό από οδηγία μου είναι κατανοητή, αλλά, υπάρχει πάντα ένα μεγάλο αλλά, έχουμε λοιπόν ε, προβλήματα μπροστά μας. Τι σημαίνει λοιπόν ε, αυτή η προσέγγιση πακέτο οδηγία, κανονισμός. Τα βλέπουμε μαζί και τα δύο. Είναι πραγματικά πακέτο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Κοινό μυστικό πιστεύω είναι ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δεν θα ήθελαν και τόσο πολύ αυτή την οδηγία για την εφαρμογή της νομοθεσίας Θα προτιμούσα να μην υπάρξει κανένα νομοθέτημα για αυτό το ζήτημα ως κοινοβούλιο. Πρέπει να δούμε προσεκτικά πώς θα αντιδράσουμε εάν τελικά το Συμβούλιο δεν προωθήσει την οδηγία όπως θα θέλαμε. Ε, λοιπόν τώρα, Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Κυρία Ιντφέλντ, έτσι θα το βλέπατε. Η Ιρλανδική Προεδρία λήγει σε 1,5 μήνα, έτσι δεν είναι. Ο ούπο. Ο κύριος Δρούτσας, ξέρετε, ήταν ε, ε, ε, Υπουργός Εξωτερικών και αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών με το 2011. Γι' αυτό αναφέρθηκε και στην πείρα του από τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου. Κυρία Εντφέλτ. Ναι. Νομίζω ότι καλό θα ήταν ε, να είχαν τελειώσει όλα υπό την ελληνική προεδρία. Έτσι λέω πάντα στους Έλληνες, μη θυμώνετε αλλά εκδικηθείτε. Είναι θέμα και πολιτικής ηγεσία. Υπάρχουν μερικά στοιχεία που είναι πιο σημαντικά από άλλα βέβαια. Μερικοί παραπονούνται για την έντονη πίεση των επιχειρήσεων, αλλά εμείς δεν παραπονούμαστε για τέτοιες ποιώσεις, αφού είμαστε ανεξάρτητοι, τουλάχιστον έτσι θεωρούμαστε, και μπορούμε να εκπροσωπήσουμε οποιοδήποτε συμφέρον θέλουμε, αφού θα είμαστε υπόλογοι προς τις εκλογές μας. Απ' την άλλη μεριά όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το lobbying, η πίεση, γίνεται με πολύ οργανωμένο τρόπο και, πολύ χρημα... και με υψηλή χρηματοδότηση. Αλλά και οι κυβερνήσεις μας πιέζουν, ακόμη και στην φάση της συγγραφής, της σύνταξης. Και αυτό δεν είναι πολύ αρμόζον. Ενώ σε άλλα θέματα, για άλλα θέματα, βλέπουμε πολύ περισσότερη συζήτηση από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και κοινωνία των πολιτών. Εδώ ναι με ορισμένε συμμετέσχων αλλά με λιγότερο ορατό τρόπο από ό,τι για άλλα θέματα. Όσο για τους πολίτες θυμάμαι την εξέγερση στο ίντερνετ κατά του άκτα που πέτυχε τελικά εμένα εγώ παίρνω συνέχεια ηλεκτρονικά μηνύματα κατά της κακομεταχείρισης των αδεσπότων σκύλων. Γιατί όμως οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται μαζικά και για το θέμα αυτό, γιατί δεν απευθύνονται στους ευρωβουλευτές τους, γιατί δεν το συζητάνε σε εθνικό επίπεδο. Ίσως γιατί το θέμα είναι τεχνικό. Είναι όμως πολύ σημαντικό να βγει και δημόσια προς τα έξω να συζητηθεί δημόσια. Και τέλος, και ίσως αυτό να μην σας αρέσει, να μην ξεχνάμε ότι μιλήσαμε πολλές φορές για θέμα προστασίας δεδομένων, αλλά τελικά, αντίθετα από τον εισηγητή μας εδώ, Kid. Εγώ δεν είμαι η ίδια Whiz Kid, δεν ασχολούμαι συνεχώς δηλαδή με τα ηλεκτρονικά, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όλοι τα πάντα για αυτές τις λεπτομέρειες και έτσι μπορούν πιο εύκολα να επηρεαστούν οι βουλευτές από λόμπι, επειδή δεν έχουν πλήρη γνώση. Μήπως θέλουν οι δημοσιογράφοι να θέσουν δύο-τρία τελευταία ερωτήματα πριν ακούσουμε τα συμπεράσματα ή κανένα σχόλιο. Ορίστε. Από εσθονικό, εκπρόσωπος εσθονικού τύπου. Τι μελέτη αντικτύπου προβλέπετε. Γιατί η αρχική μελέτη αντικτύπου ή αξιολόγηση αγνόησε αγνοήθηκε. Οι υπολογισμοί ότι 2,3 δισεκατομμύρια θα εξοικονομούνταν σε τι βασίζονται. Το κόστος που προβλέπεται για τους υπόλοιπους παράγοντες εκτός των επιχειρήσεων έχουν, έχει εκτιμηθεί δεόντως. Αυτό ρωτώ, αυτό, αυτό. Κύριε Άλμπρεχτ, δεν μπορώ να κρίνω πώς γίνονται οι μελέτες αντικτύπου της Κομισιόν. Ξέρω όμως γιατί είμαι και στην Νομική Επιτροπή όπου καθορίζουμε τους κανόνες για την εφαρμογή τους ότι υπάρχουν κανόνες. Ότι δεν γίνονται αυθαίρετα Δεν είναι δηλαδή κάτι που απλώς είναι θέμα ευχολογίου. Παρόλα αυτά, αν γίνει νομοτύπος μία αξιολόγηση ή μελέτη αντικτύπου, δεν σημαίνει ότι είναι και τελείως αντικειμενικό. Μπορεί να έχει επηρεαστεί από ορισμένους ερευνητές που έχουν συγκεκριμένες ιδέες. Είναι μία κατεύθυνση και η μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν έδειξε τα ωφέλη που θα είχε αυτή η νομοθεσία καθώς και μερικά προβληματάκια αλλά έγιναν και άλλες μελέτες η αξιολόγηση λοιπόν της Κομισιόν μου φάνηκε η πιο αντικειμενική από όλες τις μελέτες που έγιναν διάβασα μία μελέτη από το εμπορικό επιμελητήριο των ΗΠΑ που λέει ότι αν γίνει σεβαστό το δικαίωμα στη λύθη ή στη διαγραφή που ήδη ισχύει τότε λέει θα χαθούν 4.000 ευρώ ανά νοικοκυριό και ανά χρόνο στην Ευρώπη πράγμα το οποίο θα σήμαινε 500 δισεκατομμύρια το χρόνο Ενώ μιλάμε για κάτι που ήδη υπάρχει το δικαίωμα στη διαγραφή. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ούτε βασίζονται σε καμία αντικειμενική πληροφόρηση. Αν τυχόν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε το κύριο θέμα δεν θα έπρεπε να ήταν πια η κρίση, αλλά μόνο η προστασία των δεδομένων. Υπάρχει πολλή προπαγάνδα που ακούγεται, την οποία δεν πρέπει να τη θεωρούμε αντικειμενική όταν γνωρίζουμε τα πράγματα. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε το ίδιο το κείμενο και τις νομικές του ρήτρε που ήδη ισχύουν και επαναλαμβάνονται στον κανονισμό. Έτσι θα δούμε ότι τα περισσότερα θέματα που συζητούμε συνέχεια είναι αυτά που ήδη ίσχυαν από την οδηγία και άρα έχουν ήδη μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. Το βασικό είναι αυτό, ότι είναι η ίδια ερμηνεία. Απλώς θα πρόκειται για ένα ενιαίο νόμο και όχι 27 διαφορετικούς. Αυτό έχω να απαντήσω. Δεν αναμένω αυτές οι τέτοιου είδους αξιολογήσεις και άλλες μελέτες να είναι πάντοτε 100% σωστές. Αλλά βοηθάνε. Ιδίω η αξιολόγηση της Κομισιόν. Που είναι και ε, υποχρεωτικό να γίνει. Κυρία Ίντφελτ, είπατε λίγο, λίγο, ούτε λίγο. Όχι, όχι, καλά. Κύριε Τρούτσα, ούτε, καλά. Πρέπει να φύγετε μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Έχουμε παρόντες δύο εισηγητές. Υπάρχει κάποιο τελευταίο σχόλιο ή ερώτηση. Παρακαλώ. Είπατε το δικαίωμα διαγραφής είναι στον ευρωπαϊκό και εθνικό νόμο ήδη από το 95-96 Χθες ωστόσο αναφέρθηκε η περίπτωση ενός ε, Γερμανού ή Αυστριακού που έψαξε τα στοιχεία του στο facebook και είδε ότι ακόμη και αυτά τα οποία είχαν διαγραφεί στο facebook κάπου είχαν αποθηκευθεί. Προπέτασμα καπνού είναι όλα αυτά που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κάνουν ό,τι θέλουν με τα προσωπικά δεδομένα. τι έννοια έχει ένα νέο δικαίωμα που κανείς δεν ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει. Γιατί να μην υπάρχει απλώς υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τον α, β και γ τρόπο τα δεδομένα. Τον Ιαπούτσικ δουλεύω για το Αυστριακό Γραφείο των Αυστριακών Συνδικάτων. Για τον κανονισμό, ένα θέμα που δεν καλύφθηκε πολύ είναι τα συμβόλαια απασχόλησης. Ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή σήμερα το πρωί. Πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το τεράστιο όφελος για τους εργαζόμενους με τον νέο κανονισμό. Πώς βελτιώνεται για την προστασία δεδομένων των εργαζομένων. Και ακόμη, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει παραγγείλει μια μελέτη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Δημοσιεύθηκε πριν από δύο εβδομάδες και ένα πόρισμα περιέχει σαφή σύσταση προς την Επιτροπή να αντικατασταθούν τα ελάχιστα στάνταρ του άρθρου 82 με μια οδηγία για τα συμβόλαια απασχόλησης. δεν θα ήταν σκόπιμο να προωθήσετε αυτό το αίτημα. Το ερώτημα του κύριου Μιχαλ Μότσεκ, παρακαλώ. Νομίζω ότι πιο αρμόδιος είναι ο Γιάνν Άλμπρεχτ για το δικαίωμα λήθης. Αλλά να σας πω την άποψή μου. Από την αρχή το έχουμε συζητήσει πολύ το θέμα αυτό συζητώντας με τους ειδήμονες, τους πραγματικούς ειδήμονες, θέτω το ερώτημα, είναι εφικτό κάτι τέτοιο στην πράξη. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα στοιχεία σας θα διαγραφούν από το ίντερνετ. Και κυρίως μου απαντήσανε όχι. Από τεχνική άποψη ποτέ δεν μπορεί να είσαι απόλυτα σίγουρος. Άρα μάλλον έχετε δίκιο. Γιατί να εισαγάγουμε διατάξεις αν δεν μπορούμε να είμαστε πραγματικά σίγουροι ότι θα εφαρμοστούν πλήρως. Δεν είναι και καινούριο αυτό το θέμα. Ήδη είναι στην ισχύουσα οδηγία. Όμως νομίζω ότι είναι καλό να έχει αυτές τις δυνατότητες ο πολίτης και να δούμε πώς ε, σε τελευταία ανάλυση θα εφαρμοστούν αυτές οι δυνατότητες. Και αν δεν είμαστε σίγουροι ότι θα εφαρμοστεί πλήρως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να το έχουμε καθόλου, γιατί η τεχνολογία προοδεύει. Μπορεί να υπάρξουν ε, καλύτερες λύσεις στο μέλλον. Παρακαλώ κύριε Άλμπερτ για το ίδιο ερώτημα. Το δικαίωμα διαγραφής είναι νομικά θεσμευτικό ήδη με την ισχύουσα οδηγία εφαρμόζεται από την εθνική νομοθεσία υπάρχει στην εθνική νομοθεσία εδώ και 18 χρόνια και αν δεν το εφαρμόζουν οι εταιρείε και οι επιχειρήσεις είναι παράνομο. Τελεία. Πολλές επιχειρήσεις στην Ευρώπη σέβονται και εφαρμόζουν τους εθνικούς κανόνες προστασίας δεδομένων και άρα έχουν έλλειμμα ανταγωνιστικότητας έναντι αυτών που δεν τηρούν πλήρως αυτούς τους κανόνες. Προφανώς λοιπόν χρειάζεται καλύτερη αστυνόμευση της εφαρμογής των διατάξεων αυτών εάν δούμε αυτά τα οποία υπόθηκαν ε, για τον Μαξ Χέμπ από την Αυστρία. Έστειλε στο facebook έτοιμα να διαγραφούν τα στοιχεία του και δεν διαγράφησαν. Πρόβλημα, πρόβλημα, προφανές πρόβλημα. Δεν είναι η μόνη περίπτωση. Διάφορα άτομα έχουν προβλήματα όταν προσπαθούν να εφαρμόσουν τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι μόνο προβλήματα ασφάλειας ή τεχνικά. Είναι θεμελιώδη δικαιώματα αυτά. Πρέπει να το τονίσουμε. Τα θεμελιώδη δικαιώματά μας δεν απειλούνται μόνο από αυταρχικά καθεστώτα, αλλά και από άλλους Ακόμη και ο επικεφαλής ε, του Google το έγραψε πρόσφατα στο βιβλίο του «Ο διασυνδεδεμένος κόσμος». Ε, τα δεδομένα... Α, κάτι ακόμη, όχι, κάτι ακόμη. Είπατε, γιατί εφόσον δεν ε, εφαρμόζεται το ισχύον δίκαιο χρειάζονται περαιτέρω διατάξεις. Τι σχέση έχει αυτό. Θέλουμε να εφαρμόσουμε τον ισχύοντα νόμο. Βεβαίω, να βελτιώσουμε την εφαρμογή του, το θέλουμε. Και δεύτερον, γιατί όλο και περισσότερες πληροφορίε δημοσιοποιούνται αντί να περιέχονται σε κάποιο σύστημα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα εφαρμογής ε, όταν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία είναι σημαντικό, αλλά το θέμα της διαγραφής είναι διαφορετικό. Τεχνικά μπορούν να διαγραφούν τα στοιχεία. εκτός αν υπάρχουν ε, σε κάποιους τομείς ε, ανησυχίες. Γιατί να μην μπορούμε να πούμε οι επιχειρήσεις πρέπει αμέσως να διαγράφουν τα δεδομένα δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα ούτε να τα δώσουν σε άλλες επιχειρήσεις ούτε να τα αποθηκεύσουν. Μα υπάρχει αυτό στην νομοθεσία όπως λέει η νομοθεσία, ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να ασφαλή, αλλά παρόλα αυτά κάποιοι, τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι ασφαλή λέει ο νόμος, αλλά κάποιοι φτιάχνουν αυτοκίνητα που δεν είναι επαρκώς ασφαλή. Ο νόμος υπάρχει. Είναι θέμα εφαρμογή του. Ακριβώς σε αυτό το σημείο, ως νομοθέτες, θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Τώρα οι προσδοκίες των εργαζομένων. Μέχρι τούδε δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων των εργαζομένων. Η οδηγία του 95 εφαρμόζεται και για τα στοιχεία απασχόλησης. Τα στοιχεία αυτά υπάγονται στο ίδιο σύστημα με όλα τα άλλα προσωπικά δεδομένα σε κάποια κράτη-μέλη. Έχει γίνει συζήτηση για να υπάρξουν επιπλέον νόμοι για την προστασία των δεδομένων απασχόλησης. Αλλά δεν έχω υπόψη μου χώρες που να έχουν εφαρμόσει νομοθεσία για προστασία των στοιχείων απασχόλησης. Έχουν γίνει συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μια τέτοια οδηγία, αλλά δεν κατέληξαν. Οπότε, η Κομισιόν δεν έχει προτείνει συμπληρωματική προστασία για τα δεδομένα αυτά στον κανονισμό. Απλώς υπάρχει δυνατότητα στο μέλλον. Θα μπορούσε μέσω κατεξιοδότηση πράξης να κάνει κάτι τέτοιο στο μέλλον και χορηγεί και στα πλαίσια του κανονισμού δυνατότητα αυτά και στα κράτη-μέλη. Εμείς ως Κοινοβούλιο λέμε ότι δεν προτιμούμε τη λύση της κατεξοδότηση πράξης, γιατί αλλιώς θα μπορούσαμε να έχουμε ένα γενικόλογο νόμο και μετά να αναθέσουμε στην Κομισιόν ε, να τα ρυθμίσει όλα μέσω τέτοιων πράξεων. Αν θέλει η Κομισιόν, μπορείτε να τα συμπεριλάβει τώρα τα θέματα αυτά στον κανονισμό, είτε να προτείνει χωριστή οδηγία. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται αναλυτικοί κανόνες για την προστασία αυτών των στοιχείων, αλλά θα υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες και εκ των υστέρων τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να αποφασίσουν επιπλέον κανόνες. Θα υπάρχουν μερικοί λοιπόν κανόνες, τα κράτη-μέλη μπορούν να τους ενδυναμώσουν και αν εμείς ως Ευρωπαίοι νομοθέτες θέλουμε επιπλέον κανόνες, μπορούμε να τροποποιήσουμε τον κανονισμό, να προτείνουμε μια νέα οδηγία. Αλλά δεν είναι του παρόντος. Και δεν έχουμε δικαίωμα ούτως ή άλλως νομοθετικής πρωτοβουλίας. Είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να τεθεί σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον προς την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι οδεύουμε προς την ε, λήξη. Κύριε Δρούτσα, κύριε Άλμπρεχτ, θέλετε να μας πείτε μερικά επιγραμματικά, καταληκτικά λόγια, να δώσετε το όραμά σας για το μέλλον. Ο κύριος Δρούτσας, παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Έχουν υποθεί τα περισσότερο. Ένα θέμα θα ήθελα να προσθέσω που δεν είχα την ευκαιρία μέχρι τώρα να το θίξω. Είναι ένα γενικότερο σχόλιο. Πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα πετύχαμε πολύ ψηλά πρότυπα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο. Τολμώ να πω ότι σε αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος και πρωταγωνιστής. Και στόχος μας θα έπρεπε να είναι να διατηρήσουμε αυτά τα υψηλά πρότυπα και τον πρωταγωνιστικό αυτό ρόλο σφαιρικά παγκοσμίω. Αυτό το βλέπουμε και στις συνεννοήσεις μας με τους Αμερικανούς σε πολλά θέματα όπου όποτε τίθεται το θέμα της προστασίας των δεδομένων αν συγκρίνουμε τα συστήματα όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και με πολλές άλλες χώρες και υπήρους βλέπουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πετύχει πολύ ψηλά πρότυπα. Αυτός πρέπει να συνεχίσει να είναι ο στόχος μας. Ξέρουμε ότι έχουμε διαπραγματεύσεις και θα έχουμε για τις ελεύθερες συναλλαγές με τη ΣΥΠΑ και είναι γνωστό ήδη ότι θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων θα τεθούν στις διαπραγματεύσεις αυτές και θα ασκηθεί πίεση. Ιδιαίτερα εφόσον μας προκαλεί και η οικονομική κρίση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Τα επιχειρήματα λοιπόν για δημιουργία θέσεων απασχόλησης κλπ. κλπ θα ακουστούν και θα ξανακουστούν για την ανταγωνιστικότητα και τα λοιπά. Είναι σημαντικά θέματα, αλλά δεν πρέπει να θυσιάσουμε τα υψηλά πρότυπα που έχουμε πετύχει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο βωμό της αντιμετώπισης της κρίσης. Και επειδή είναι επίκαιρο θέμα, και την επόμενη εβδομάδα θα το θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στον ενεργειακό τομέα η ίδια επιχειρηματολογία ακούγεται. Υπάρχει κρίση και γι' αυτό να δούμε πώς θα πετύχουμε φτηνότερη ενέργεια. Ναι, σημαντικό πράγμα η φτηνή ενέργεια, αλλά πρέπει να είναι φτηνή και καθαρή. Να μην ξεχάσουμε το μέλλον και το ίδιο ισχύει και για την προστασία των δεδομένων. Το λέω γιατί προβλέπω άσκηση τεραστίων πιέσεων και προς και από το Συμβούλιο. Λόγω της σύμπτωσης αυτής, ότι υπάρχει δηλαδή οικονομική κρίση με τις διαπραγματεύσεις της ΣΥΠΑ για τις ελεύθερες συναλλαγές και ούτω καθεξής, προβλέπω πολύ υψηλή πίεση στο Συμβούλιο και από το Συμβούλιο και ίσως να εκφραστεί ο πειρασμός να μειώσουμε τα πρότυπά μας. Οι συνάδελφοί μας λοιπόν στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις δεν πρέπει να ξεχάσουν ποιος είναι ο στόχος. Είναι τα δικαιώματα των πολιτών μας. κύριος Άλμπρεχτ. Έχετε εμπιστοσύνη στο μέλλον εσείς. Πάρα πολύ. Διότι όπως είπα και πριν όλα τα ευρωπαϊκά όργανα σαφώς αναγνώρισαν ότι υπάρχει ανάγκη για υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων. Και ξέρω ότι τεράστια πλειοψηφία του κόσμου, των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρεται για το θέμα της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Και επανειλημμένος έχω δει ότι υπάρχει ανησυχία για αυτό το θέμα, τι γίνεται με τα στοιχεία μου, τι τα κάνουν, τι δικαιώματα έχω όταν μπαίνω σε ένα κοινωνικό δίκτυο κλπ. κλπ. Τους ενδιαφέρει το θέμα. Πολλοί βέβαια θα ήθελαν να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά ιδιαίτερα ως νέος πολιτικός συναντώ πολλούς ιδιαίτερα νεότερους που πολύ πιο συχνά από τους μεγαλύτερους βάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα στο ίντερνετ κλπ. Και ανησυχούν όλοι, ενδιαφέρονται. Και μου λένε, σας παρακαλούμε, σεβαστείτε τον ιδιωτικό χαρακτήρα των δεδομένων αυτών, γιατί χρειαζόμαστε τους κανόνες προστασίας. Και δεν μπορώ να προβλέψω κακό αποτέλεσμα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αν τον κανονισμό αυτόν τον εγκρίνουμε χωρίς να αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα όλων των πολιτών, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της θα απολέσει εμπιστοσύνη, αξιοπιστία στα μάτια των πολιτών. Γιατί εδώ προσπαθούμε να δείξουμε ότι η Ένωση υπάρχει για να μας προστατεύει, ας πούμε, ως προς τα προσωπικά δεδομένα, για τα θεμελιώδη μας δικαιώματα και άρα πρέπει να θεσπίζει κανόνες και κατά τη συμπεριφορά ορισμένων μεγάλων εταιριών που δεν σέβονται πάντοτε τα ισχύοντα. Αν δεν το κάνουμε αυτό θα χαθεί η εμπιστοσύνη και δεν πιστεύω να θελήσει κανείς να αναλάβει αυτόν τον κίνδυνο. Γι' αυτό έχω εμπιστοσύνη ότι πολύ σύντομα θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Και θα φανεί έτσι ότι μπορούν να καθοριστούν κανόνες και στις Ηνωμένε Πολιτείες όπου λέμε ότι διαφωνούν και εκεί οι πολίτες έχουν τις ίδιες ανησυχίες και ενδιαφέροντα και στην Νότια Αφρική και στην Ιαπωνία παντού. Τις ίδιες ανησυχίες και ενδιαφέροντα έχει ο κόσμος και θα το θίξει, θα φανεί ακόμη και για την ψηφιακή αγορά και σε πλαίσια οικονομικής κρίσης θα φανεί ότι μπορούν να τεθούν κανόνες ως προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία της κοινωνίας και της αγοράς. Και είναι σημαντικό να δηλώσουμε ότι κανείς δεν θέλει να απαγορέψει τίποτα από κανέναν, απλώς μιλάμε για προϋποθέσεις σωστής κοινή διαβίωσης και εργασίας. Γι' αυτό ας πούμε η Επίτροπος Ρέντινγκ που είναι συντηρητική και εγώ ένας πράσινος ακτιβιστής συμφωνούμε σε τέτοιο βαθμό. Μάλιστα. Και αυτά ένα χρόνο πριν τις επόμενες ευρωεκλογές. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ όλους τους συναδέλφους που συμμετέσχουν στη συζήτηση, τους δημοσιογράφους που σχολίασαν, τους ε, διερμηνείς, merci μποκού, και τέλος τη γραμματεία μας για την πολύτιμη βοήθεια που μας παρέσχε για τη διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου. Μία λεπτομέρεια σημαντική, υπάρχει μια δεξίωση αμέσως μετά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στον πέμπτο όροφο